Ja, ich eröffne die Sitzung von heute Mittag. Nachdem wir heute Morgen alle so zahlreich waren, war es uns klar, dass wir heute Mittag. Αρχίζει η συνεδρίαση. Weil das Thema auch nicht unbedingt jedermanns Thema ist. Alle Football Girls and Boys sind. Έχουμε ένα θέμα το οποίο βέβαια μπορεί να μην απασχολεί του πάντε, αλλά βλέπω δεν έχουν έρθει ούτε οι άντρε που θα έπρεπε να ενδιαφέρονται για την παλίτσα. Ελπίζω να έρθει κανένα. Τέλο πάντων, έτσι είναι αυτά. Μα κάνει κανεί ακρόαση λίγο πριν από τα Χριστούγεννα. Ε, έτσι είναι. Τα παθήματα γίνονται μαθήματα. Στο μέλλον δεν θα τα ξανακάνουμε. Δεν βοηθάει και τους... τι να πω και στους τρεις προσκεκλημένους μας. Τόσο οι άνθρωποι που έχετε πάντως θα ακούσουν με μεγάλη προσοχή. Γνωρίζετε, γι' αυτό είστε και εδώ πέρα άλλωστε σήμερα, πως ε, από τη Λισαβόνα και μετά έχουμε κάποιες αρμοδιότητες για τον αθλητισμό και βεβαίω υπάρχει και λευκή βίβλος για τον αθλητισμό που εξεργάστηκε ο Φίσες αλλά δεν έχουμε και μεγάλες προσδοκίες ε, αυτό το οποίο αναμένουμε είναι να έχουμε κάποιους κανόνες ε, για τον αθλητισμό, το, το ποδόσφαιρο, έτσι, ευρία ταινία και ζητήματα ανταγωνισμού, στοιχήματος εκεί όπου είχαμε κάποιες, ε, πώς να το πω, ατασταλίες. Αυτά προσπαθούμε, δυστυχώς. Ένας εμπειρογνώμονας από την UEFA μας είπε σήμερα το πρωί ότι δεν θα έρθει κιόλας για λόγους σημαντικούς. Μου είπε Επαγγελματικού λόγους δεν μου είπε τι. Ε, φαντάζομαι ο κύριος Πλατινή τον ήθελε επιγόντω. Αλλά από τους ε, τρεις παρόντες, τον κύριο Μίταγ, ε, Άντρισεν και Γκάλικ, Ολλανδός, Γερμανός και Δανός δηλαδή, Είμαστε και εμείς εδώ πέρα, εγώ είμαι Γερμανίδα, ο κύριος Λόκεγκαρτ είναι βεβαίως από την Δανία. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε θα μας πείτε. Ε, με το Πανεπιστήμιο της Κολονίας βεβαίως έχουμε σχέσεις εδώ και χρόνια. Όταν είχα γράψει την πρώτη μου έκθεση τότε το 1996 ε, είχα τις πρώτες επαφές με το Πανεπιστήμιο της Κολονίας. Είναι και εδώ πέρα και ο κύριος Γκαλίκο από το κλάδο επιχειρήσεων της Europol ε, στη Χάγη. Κύριος Γκάρλικ και ελπίζω να καλύψουμε τα ζητήματα. πάντων, δεν θέλω να μιλήσω περισσότερα. Θα δώσω, το, λόγο σε εσά να μα παρουσιάσετε τα προβλήματα. Ε, όπως ε, τα βλέπετε εσείς ως ειδικοί. Και μετά θα έχουμε δυνατότητα να συζητήσουμε. Επειδή δεν έχει έρθει και ένας ειδικό, έχουμε περισσότερο χρόνο, αλλά μην το παρακάνουμε. Και όταν τελειώσετε θα τελειώσει και η συνεδρίαση. Λοιπόν, ποιο θέλει να ξεκινήσει. Κύριε Γκάρλικ, έχετε το λόγο. Αγγλικά θα μιλήσετε, ναι. Τα-τα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ σήμερα σε αυτή την πάρα πολύ σημαντική ακρόαση και πραγματικά σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Ονομάζομαι Νίκ Γκάλικ και πήρα μέρος σε, αυτή την, σε αυτό το εγχείρημα της Europol που άρχισε δύο χρόνια πριν ε, και προηγουμένως δούλευα στην Intelligence Service στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το θέμα των στοιχημάτων και των καταχρήσεων των αστασταλιών που γίνονται δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Ε, υπήρξε το σκάνδαλο του Αμερικανικού baseball τον περασμένο αιώνα ε, και πολύ πιο πρόσφατες ε, περιπτώσεις στη Γαλλία και στην Ιταλία. Υπήρξαν πολλές ε, περιπτώσεις επίσης ατασταλιών και στο κρίκετ. Το έγκλημα είναι ένα καθολικό φαινόμενο και ε, το θέμα των στοιχημάτων καθιστά πιθανό για μια ομάδα εγκληματιών από το ένα μέρος του κόσμου να στοιχηματίσουν πάνω σε ένα μικρό αθλητικό γεγονός και να καθορίσουν την έκβαση του αγώνα. Αυτό συμβαίνει και αυτό συνέβη και σε περίπτωση μας πολλές φορές τεράστια ποσά σε ρευστό χρήμα ανταλλάσσονται κάτω από το τραπέζι και ε, τεράστια στοιχήματα κατατίθενται. Οπότε ε, πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση και πώς θα αντιμετωπίσουμε τα, τους διάφορους ιστότοπους στο διαδίκτυο που, όπου καταγράφονται στοιχήματα, όπου οι άνθρωποι στοιχηματίζουν ηλεκτρονικά. Ε, υπάρχει και το θέμα των αγώνων ποδοσφαίρου ε, και οι ε, αυτοί που βάζουν τα στοιχήματα αντιμετωπίζουν μια και δημιουργούν μια αφόρητη κατάσταση ε, και αυτό φαίνεται να παραχαράσει το πνεύμα του αθλητισμού και να χρησιμοποιεί το αθλητισμός για τα στοιχήματα. Είναι κάτι το οποίο επίσης φουντώνει στην Ασία και σε πάρα πολλά εκατομμύρια νομίμων στοιχημάτων υπάρχουν πάντα αυτοί που θέλουν να παραχαράξουν τα στοιχήματα και να ανατρέψουν την έκβαση των αγώνων. Ε, υπήρξε ε, ε, ένα τεράστιο, είναι μια τεράστια εισοδηματική πηγή μέσα από τα στοιχήματα τα τελευταία χρόνια για πολλούς και ένα, μια ομάδα κρατών μελών τα τελευταία χρόνια άρχισε, ξεκίνησε μια έρευνα για να ε, δει τι γίνεται στον τομέα των στοιχημάτων και από μόνο σε πολλές περιπτώσεις σε, διάφορες, σε διάφορα κράτη-μέλη ε, και απευθύνθηκε στις αρχές επιβολής του νόμου και στις κρατικές αρχές. Ο καταλληλότερος τρόπος ε, γι' αυτό ήταν να του ζητήσει να πάρουν μέρος στην έρευνα. Έτσι δημιουργήθηκαν ομάδες έρευνας, ε, ε, συνήψαν μια συμφωνία και με τα κράτη-μέλη και τις αρμόδιες αρχές άρχισαν να ασχολούνται με το θέμα των στοιχημάτων. Ο στόχος του όλου εγχειρήματος ήταν να ερευνήσουν συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ξεκινώντας μπορεί κανείς να πει ότι συνδέεται το θέμα των στοιχημάτων με διάφορες χώρες της Ευρώπης και εκτός Ευρώπης ε, και παραχαράσει τους κανόνες του ανταγωνισμού. Έχουμε τα παιχνίδια ύστερα στο ίντερνετ, τα στοιχήματα στο ίντερνετ και τα οποία καταλήγουν στη διαφθορά των παιχτών και στη, διαφορά, στη διαφθορά των προπονητών και των οργανωτών. Και είναι πια μέρος του οργανωμένου εγκλήματος το στοίχημα. Πρέπει λοιπόν ε, να καταλάβουμε ότι πολλές φορές ε, το έγκλημα παίρνει μεγάλες διαστάσεις γιατί θέλουν πραγματικά να αλλάξουν την έκβαση του αγώνα και υπάρχει τεράστια απώλεια αν γίνει κάτι διαφορετικό στις, ε, στα χρήματα που παίρνουν για, για, την, για τον καθορισμό της έκβασης του αγώνα. Οπότε είναι πάρα πολύ μεγάλες και οι απώλειες και τα κέρδη και ο κίνδυνος είναι τεράστιος και μπορούμε να πούμε ότι σε πάρα πολλούς άλλους τομείς του οργανωμένου εγκλήματος τα κέρδη δεν είναι τόσο ισχυρά. Τον Σεπτέμβριο του 2011 ε, έγιναν ορισμένες συλλήψεις και μάλιστα παικτών διεθνών ε, και Ιταλών πολύ γνωστών παικτών έγινε μια έρευνα ε, η οποία αποκάλυψε πάρα πολλά σκάνδαλα και πάρα πολλά μυστικά και υπάρχει κάθε συμφέρον να συνεχιστεί αυτή η έρευνα. Βεβαίως ε, υπήρξαν ε, αρχικά οι υποψίες που οδήγησαν τους όσους ασκούσαν την έρευνα στον, στα άτομα ε, που είχαν κάνει τις ατασταλίες πρέπει να πούμε ότι η επιτυχία αυτής της σημερινής έρευνας ήταν ανέλπιστη και το ποδόσφαιρο πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι ο μόνος τομέας όπου υπάρχουν ατασταλίες και υπάρχουν υπενιγμοί για χειραγώγηση και άλλων αθλημάτων όπως είναι το κρίκετ για παράδειγμα και πρέπει να γίνουν περισσότερες έρευνες για να ληφθούν όλα τα στοιχεία που έχουμε σοβαρά μέχρι να καταλήξουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Οι εγκληματίες θεωρούν ότι είναι εγωιτευτική αυτή η πηγή χρηματοδότησης. Ε, είναι ένα χαμηλό επίπεδο σε σχέση ε, με άλλα ε, εγκληματικά επίπεδα, αλλά ωστόσο αν αρχίσουν να καταδικάζονται ορισμένοι εγκληματίες θα απειληθεί όλο το σωιστός του οργανωμένου εγκλήματος για τα στοιχήματα. Έχουμε δύο μεγάλα γεγονότα. Φέτος το καλοκαίρι οι Σκανδιναβοί ε, οργανώνουν αγώνες κατά τη διάρκεια του θέρους. So... καλοκαίρι όταν δεν υπάρχουν τα άλλα πρωταθλήματα για να μπορούν να συνεχίσουν να στοιχηματίζουν και αυτό ε, κάνει πάρα πολύ ελκυστικό το εγχείρημά τους και είναι πολύ καλό πληρωμένο. Ε, πρέπει να πούμε, ε, δεν πρέπει να πούμε ότι οι χειραγωγήσεις βρίσκονται μόνο σε αυτό το τομέα. Ε, υπάρχουν επίσης και πάρα πολλοί ηθήνοντες που ασχολούνται με τον αθλητισμό οι οποίοι είναι διεφθαρμένοι ε, και οι οποίοι είναι θύματα του οργανωμένου εγκλήματος. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει να εξεταστεί πάρα πολύ σοβαρά για να μπορέσουμε να έχουμε τη διαβεβαίωση ότι θα υπάρχει κάποια κεραιότητα ε, σε όλες αυτές τις αρχές. Οι εισηγήσει που μας δόθηκαν σε διάφορα μέτρα ε, μας έδωσαν τη δυνατότητα να ε, ερευνήσουμε πάνω στα στοιχήματα. Είχαμε ανώνυμες πληροφορίες σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες. Δημιουργήθηκε επίσης, είναι σημαντικό, ένα περιβάλλον από τους παίκτες οι οποίοι ήδη είχαν κατηγορηθεί για τα σταλίες και βέβαια το μόνο αποτέλεσμα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να δημιουργηθεί ένα επίπεδο υψηλού φόβου ε, και να μην ε, μπορούν οι αρχές να προχωρήσουν. Τελικά τα, παιχνίδια των οποίων η έκβαση είναι προκαθορισμένη ε, είναι το αντικείμενο της έρευνας, της αρχικής έρευνας. Εμείς, εγώ δεν ξέρω, θα ήθελα να ακούσω και οι άλλοι συνάδελφοι τι λένε για να μπορέσουν να συνεχίσουν τη συζήτηση πάνω σε αυτές τις πληροφορίες που έχουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα δώσω τον λόγο στον κύριο Μίταγκ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να επικεντρωθώ στον τομέα του Financial Fair Play, ένα θέμα το οποίο συζητιέται συχνά στα ΜΜΕ ως επανάσταση στον αθλητισμό, αλλά βεβαίως αυτοί οι οποίοι μιλάνε για το θέμα δεν ξέρουν συχνά περί τίνο ε, πρόκειται. Θα αναφερθώ λοιπόν πρώτα απ' όλα στο πλαίσιο, μετά στο financial fair play και μετά στα όρια και τις δυνατότητες του. Πρώτα απ' όλα, σημασία έχουν οι οικονομικές εξελίξεις για το πλαίσιο έχουμε μια τεράστια αύξηση του τζίρου κατά 9,1% μεταξύ 2006 και 2010 στα 12,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Βεβαίως τα περισσότερα λεφτά κινούνται στα πέντε πιο μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Βεβαίως αυξάνονται και τα χρέη, όπως ξέρετε η Βαλένσια έχει πάνω από 5 δισεκατομμύρια χρέη και βεβαίως συνολικά τα κορυφαία πρωταθλήματα είχαν, παραδείγματος χάρη το 2009, 1,18 δισεκατομμύρια ευρώ απώλειες και 1,6 δισεκατομμύρια το 2010. Και αυτό οφείλεται βέβαια πάρα, πάρα πολύ ψηλά ποσά για τις μεταγραφές. Αν δούμε λοιπόν την ε, σημασία του ε, επαγγελματικού ποδοσφαίρου μόνο στην Γερμανία. Μιλάμε για μια δημιουργία πλούτου 5 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα οποία 1,5 δισεκατομμύριο πάει στο κράτος υπομορφή φόρων. Οπότε βλέπουμε τι σημασία έχει ακριβώς η ρύθμιση ε, του ποδοσφαίρου. Ήδη αναφέρθηκε αυτό το οποίο είχε συζητηθεί η για ένα πλαφόν το οποίο βεβαίως δεν μπόρεσε να περάσει. Η αδειοδότηση μέσω της ε, UEFA που ξεκίνησε από το 2004-2005 ορίζει έναν ελάχιστο κατάλογο αλλά βέβαια δεν έχει τις ε, δυνατότητες ελέγχου η UEFA και πρέπει να λεφθούν υπόψη και οι εθνικές ιδιαιτερότητες ε, βεβαίως ιδιαίτερο ρόλο παίζει η Ισπανία που είναι μεγάλο πρωτάθλημα και δεν υπάρχει εθνικό σύστημα αδειοδότησης η UEFA ζήτησε λοιπόν άδειε από όλε τι ομάδε. Χαρακτηριστικά παραδείγματα μεγάλων ομάδων ήταν η Μαγιόρκα και η Πόρτσμουθ, οι οποίε δεν είχαν ζητήσει άδεια και έτσι άρα είχαμε πάρα πολλέ ε, διαφορέ και αυτό σημαίνει στρέβλωση του ανταγωνισμού καθώ είναι τελείω διαφορετικά τα μοντέλα των ευρωπαϊκών ομάδων. Και άρα φτάνω στο αποφασιστικό πώ έχει η διαδικασία αδειοδότηση σε σχέση με το Financial Fair Play. Σημαντικό είναι λοιπόν το ότι ο ρόλος και η είσοδος των επενδυτών στον χώρο δεν ρυθμίζεται με τρόπο ενιαίο και βεβαίως ε, υπάρχουν έτσι μεγάλες ανισότητες που προκύπτουν από αυτό. Η UEFA λοιπόν όρισε ένα σώμα που θα αναπτύξει υποτίθετο Financial Fair Play και εκεί πέρα συμμετέχει η ίδια η Ένωση ε, Ενώσεων ε, Ποδοσφαίρου για το πώς θα μπορέσει να, ληφθεί, να γίνει καλύτερα η απόφαση αδειοδότησεων ομάδων. Αυτό έγινε το 2010. Βεβαίω, όλο ο οργανισμό περιλαμβάνει 74 άρθρα σε 99 σελίδε. Ε, εν τω μεταξύ, ξεκίνησε η διαδικασία. Υπάρχει ένα ελεγκτικό συνέδριο με τον Ζαν Λουκ και ένα δικαστήριο αθλητικό της ΟΕΦΑ με επικεφαλή σε έναν πρώην δικαστή του 10. Βεβαίω όλα αυτά έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία, αλλά τι σημαίνει, ισχύουν μόνο για τι ομάδε που παίζουν στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Γίνεται η διάκριση μεταξύ σημαντικών και μη σημαντικών δαπανών ε, και βεβαίω έχουμε τι λειτουργικέ δαπάνε ο πυρήνας δηλαδή αυτού του κανονισμού οφείλεται στο ότι τα έξοδα θα πρέπει να είναι μέχρι το ύψος των ε, εσόδων σε μια καθορισμένη χρονική περίοδο. Επίσης θα πρέπει από ό,τι λένε το 2013-2014 και 2014-2015 να υπάρξουν κάποιες μεταβατικές διατάξεις που επιτρέπεται ένα έλλειμμα 45 εκατομμυρίων ετώ, ε, ευρώ, με συγχωρείτε, και το 15-16 και το 16-17 μόνο 30 εκατομμύρια ευρώ έλλειμμα το έτος. Βεβαίως από αυτό εξαιρούνται οι επενδύσεις σε υποδομές και οι ακαδημίες για τους νέους παίκτες. Όπως είπα τώρα είμαστε στην περίοδο παρακολούθησης και μπορεί να υπάρξει και ένα συνυπολογισμό με παλαιότερες περιόδους. Για να έχει λοιπόν κάποια ε, σημασία αυτό το νόημα θα πρέπει να γίνονται ανεκτές αποκλήσεις μόνο μέχρι 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Βεβαίως σημασία έχει όπως είπαμε να προσαρμοστούν τα έξοδα στα έσοδα και να υπάρξουν και ποινές σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Βεβαίως αυτό έχει και πολιτικές πιθανώς επιπτώσεις. Δηλαδή θα μπορούσε αφενός η UEFA να κάνει κάποιες επιπλήξεις, μετά πρόστιμα, αλλά και να βγάλει ομάδες από ε, ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Βέβαια, ε, κάθε ένα από αυτά τα βήματα έχει διαφορετικές συνέπειες για τα εθνικά πρωταθλήματα. Η γερμανική Bundesliga που έχει τον κανόνα 50 συν 1 θα επηρεαστεί λιγότερο. Το αγγλικό και το γαλλικό πρωτάθλημα βεβαίως θα επηρεαστεί πολύ περισσότερο γιατί βεβαίως θα μειωθούν ε, οι μεταγραφές μέσω του λεγόμενου third party ownership. Σοβαρά προβλήματα αναμένονται στην Ισπανία όπου είναι και πολύ χρεωμένες οι ομάδες. Ποιες δυνατότητες και ποια όρια τώρα έχει το σύστημα του Financial Fair Play. Πρώτα απ' όλα οι δυνατότητες. Αφενός αναμένεται να πέσουν οι εξωφρενικές δαπάνες για μεταγραφές των προηγούμενων ε, ετών. Ήδη όπως καταγράφει η UEFA έχουμε μία μείωση κατά 36% τον Ιανουάριο του 2012 σχέση με τον Ιανουάριο του 2011. Ήδη έχουν διαπιστωθεί οι πρώτες ε, αυλεψίες από 23 συλλόγους, ε, την Πεσίκτα ε, και άλλες τουρκικές ομάδες, οι οποίες από ό,τι φαίνεται θα αποκλειστούν από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα του επομένου έτους. Και επίσης από ό,τι φαίνεται απειλείται και η Μάλαγα με τέτοιο αποκλεισμό. Βεβαίως υπάρχουν και κάποια όρια στο τι μπορεί να γίνει. Πρώτα απ' όλα το Financial Fair Play περιορίζεται μόνο σε αυτές τις ομάδες οι οποίες όπως είπα παίζουν σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Δεύτερον και επίσης ε, σημαντικών παρόλες λεπτομερείς ρυθμίσεις εξακολουθούν να υπάρχουν γκρίζες ζώνες όπως παραδείγματο χάρη επενδύσει σε υποδομή ή τα λεγόμενα πάγια έξοδα που μπορεί να τα εκμεταλλευτούν η ομάδα. Επίσης ε, το Financial Fair Play θα μπορούσε να αποτελέσει πρόσχημα για λογιστικά κόλπα, για δημιουργία θηγατρικών που θα αναλάβουν τα έξοδα κτλ. Ειδικά το ζήτημα της δημιουργικής, λογιστικής ε, και ερμηνείας κυκλοφορεί σε διάφορες συζητήσεις. Ένα παράδειγμα για το τι γίνεται παραδείγματος χάρη. Η Manchester City υπέγραψε μια συμφωνία 10 ετή ύψους 504 εκατομμυρίων ευρώ για τα δικαιώματα χρήσης ε, του ονόματός της. Ε, κάτι ανάλογο υπάρχει και με την ε, Arsenal, με το στάδιο της που έχει ονομαστεί Emirates. Αλλά εκεί πέρα είναι μόνο 126 εκατομμύρια ευρώ το αντίτιμο για 15 χρόνια. Είτε λοιπόν η Manchester City είναι πολύ καλύτερη διαπραγματευτής, είτε έχουμε μια κρυφή επιδότηση. Επίσης βεβαίως σε πολύ γνωστές ομάδες που έχουν κάποιο κύριο, ε, που εμφανίστηκαν βεβαίως τελευταία στην κορυφαία κατηγορία όπως η Manchester City ή η Paris Saint Germain ε, εμφανίζουν και αυτές ε, τεράστια ελλείμματα. Παραδείγματο χάρη, η Paris saint είχε 100 εκατομμύρια έλλειμμα το προηγούμενο καλοκαίρι και επένδυσε 147 εκατομμύρια ευρώ σε μεταγραφές το καλοκαίρι που μας πέρασε. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι σημαίνει ε, να αποκλείονται μεγάλες ομάδες από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έχουμε τη βάση ε, ενός πανευρωπαϊκού δικαίου του ανταγωνισμού σε αυτόν τον ε, τομέα θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε σε μια βραχυπρόθεσμη εξυγίανση των ομάδων και βεβαίω το ζήτημα είναι πώς θα ελεγχθεί και θα εφαρμοστεί ε, ο κανονισμός ε, αυτός για να μην δημιουργηθεί ένα τεράστιο διοικητικό πλέγμα δικηγόρων και λογιστών. Επίσης ε, το ζήτημα βεβαίως αφορά και τις κρατικές ενισχύσεις και το third party ownership και το ζήτημα των θυγατρικών όπως είπα που είναι ακόμα ανοιχτά στη συζήτηση. Τέλος, τι σχέση έχει με την Ευρωπαϊκή Ένωση το Financial Fair Play. Η Κομισιόν στήριξε τον κανονισμό αυτόν στο πλαίσιο της ανακοίνωσής της για τον αθλητισμό του 2011 που λέει χαιρετίζει την εισαγωγή μέτρων με τις οποίες ε, σκοπεύεται να βελτιωθεί το ε, οικονομικό εφαγωνίζεσθε και επενθυμίζει ταυτόχρονα πώς θα πρέπει να γίνονται σεβαστές οι αρχές της εσωτερικής αγοράς και του ανταγωνισμού. Υπήρξε λοιπόν μια εξέταση ως προς το εάν συμφωνεί με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά όσον αφορά το τι μπορεί να οριστεί ως πρόοδος εδώ πέρα, αλλά βεβαίως υπήρξε και μια κοινή δήλωση Αλμούνια και Πλατινή 13 ε, σημείων ε, τον Μάρτιο του 2012. Επίσης ε, σημαντικό είναι το ζήτημα των κρατικών ενισχύσεων με τις φοροαπαλλαγές παραδείγματος χάρη στην Ισπανία. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω κάποιες ε, παρατηρήσεις για να συνοψίσω. Οπωσδήποτε το Financial Fair Play είναι κάτι που είναι ένα βήμα σημαντικό προς σωστή κατεύθυνση και το παρακολουθεί η UEFA από το 2004 σε μια διαδικασία διαχείρισης ε, του κινδύνου. Θεωρώ πως ε, είναι σημαντικό το ότι δημιουργήθηκε και εφαρμόστηκε με τη συμμετοχή πολλών ενδιαφερομένων ε, του κλάδου, κάτι το οποίο δεν ήταν αυτονόητο, οπότε έχει αφενός πολιτική στήριξη, αλλά βεβαίως από την άλλη θα πρέπει να γίνει πιο συγκεκριμένο και χωρίς ε, μεγάλους συμβιβασμούς. Επίσης ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το εξής. Όποιος βγάζει πολλά εξακολουθεί να μπορεί να δίνει πολλά. Έτσι. Οπότε δεν ανατρέπεται το status quo των, ε, του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Οπότε το ζήτημα του ανταγωνισμού και της ανισότητας πρέπει να ληφθεί υπόψη και πρέπει να δούμε το εάν ε, το financial fair play θα πρέπει να δει τις ανισότητες οι οποίες θα εδραιωθούν με αυτόν τον τρόπο αντί να ε, μειωθούν. Επίσης θα πρέπει να συζητηθεί και πολιτικά, άρα το ζήτημα συμπληρωματικών μέτρων. το χάρη, πώς θα μπορούσε να, μεταβληθεί το ζήτημα αυτό, το σύστημα αυτό, με συγχωρείτε, σε ένα σύστημα πριν. Επίσης, Βεβαίω, ε, αποφεύγεται εδώ πέρα αυτά τα, αποφεύγεται το ζήτημα το οποίο έχει θέσει η UEFA και αφορά την λεγόμενη αλληλεγγύη μεταξύ των ομάδων. Επίση, μην ξεχνάμε πως ε, όλοι οι πρωταθλητέ του Champions League ε, πλην άγιαξ και Πόρτο είναι από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα αποκλειστικά. Έτσι και αν εξαιρέσουμε την Τζέλσι που το πήρε πέρσι, ήταν οι λεγόμενες ε, G14, οι μεγάλες 14 ομάδες της Ευρώπης. Και βεβαίως βλέπουμε πόσα, πόσα διακινήθηκαν ε, το 2011 και 2012 στο Champions League ε, από την UEFA στο πλαίσιο των μέτρων αλληλεγγύης το 2010-2011 διανεμήθηκαν 238 εκατομμύρια ευρώ. Σοβαρό ποσό, αλλά βεβαίω το ζήτημα είναι σε ποιο βαθμό αυτές οι, προβλη... οι προσεγγίσεις αναπτύσσουν το ποδόσφαιρο με έναν τρόπο, όπως είπα, αλληλέγγυο διασφαλίζοντας τον ανταγωνισμό. Εν ολίγης, μια σύσταση είναι χρήσιμη αυτή η έννοια, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να παρατηρούμε το σύστημα αυτό, να το διευκρινίσουμε δεν πρέπει ε, να το αφήσει χωρίς παρακολούθηση και η πολιτική και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει επιθέτως να το παρακολουθεί εις βάθος. Ευχαριστώ κύριε Μίταγ. Περνάμε στον τελευταίο ομιλητή, τον κύριο Γιέντς Σέγερ Άντερσεν. Έχετε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε και κύριοι. Όπως μόλις ακούσαμε, το άθλημα είναι μια βιομηχανία ε, η οποία έχει παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον. Χρειάζεται να προστατεύσουμε λοιπόν το αθλήματα από κάθε παράνομη πρακτική θα πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια η σχέση μεταξύ του αθλητικού κινήματο και του υπόλοιπου κόσμου έχει φτάσει σε ένα σταυροδρόμι. Θα ήθελα να σα συγχαρώ λοιπόν που οργανώνετε αυτή την ακρόαση και θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης για την πρόσκληση από το 1997 ασχοληθήκαμε με τις ε, θετικές αλλά και τις αρνητικές ε, επιπτώσεις ε, με το ντόπινγκ, το στήσιμο παιχνιδιών και ούτω καθεξής. Πιο συχνά διαπιστώσαμε ότι οποιαδήποτε πρόκληση αντιμετωπίζαμε η λύση εξαρτάται από κάτι το οποίο ήταν πολύ δύσκολο να ξεβρεθεί. Για, με αποτελεσματική διοίκηση και με άλλα λόγια το ένα, ε, αγωνίζεστε. Θα τονίσω το θέμα της ε, χρηστής ε, διαχείρισης στο ζήτημα των, των αθλημάτων. Το, στη Βουδαπέστη το 2011, σε έναν μαραθώνιο, ένας μικρός όμως έλαβε το μικρόφωνο και είπε ότι η διαφθορά υπάρχει παντού σε όλα τα αθλήματα και επηρεάζει σε όλα τα θέματα που επηρεάζει τις ε, εξελίξεις, ακόμα και τα τεστ ε, περί ντόπινγκ. Χωρίς τη βοήθεια του κοινού δεν πρόκειται να εξευρεθεί καμία λύση. Ζήτησε από τον αρμόδιο Ευρωπαϊκό Επίτροπο να παρέμβει. Εάν δεν συμβεί τίποτα, τότε το μέλλον θα είναι άδειλον. Αυτή η προειδοποίηση δεν προέρχεται από κάποιον ριζοσπάστη ακτιβιστή, αλλά από κάποιον ε, έμπειρο, ε, ε, τον πρόεδρο της Ουγγρικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων, τον Μαυριάν, τα λόγια του ε, ότι δεν υπάρχει μονοπόλιο στα αθλήματα και ότι η FIFA αυτή τη στιγμή ε, πραγματικά ερευνάται ενδελεχώς. Μία από τις πιο πλούσιες οργανώσεις, ε, η FIVB, για 24 χρόνια, από το 1994 στο 2008, προεδρεύεται από τον Ντακώστα του Μεξικού. Αυτό εισήγαγε δύο κανόνες. Ο πρώτος είναι ότι οποιοδήποτε σπόνσερας θα μπορούσε να εισπράττει το 10% των συμβάσεων ως προσωπικό μπόνους. Και ο δεύτερο κανόνα είναι ότι ο πρόεδρος θα έπρεπε να υπογράφει όλες τις συμβάσει. Όταν μερικοί θαραλέοι αξιωματούχοι άρχισαν να επικρίνουν τότε ο, Κώστα, ο Ακώστα πρότεινε να ληφθούν μέτρα. Η FIVB αποδέχθηκε σε μυστικά έγγραφα ότι ο Ακώστα έφυγε με ένα προσωπικό κέρδος τουλάχιστον 32 εκατομμυρίων δολαρίων. Λοιπόν, η τιμή του καθεστώτος, το τίμημα του καθεστώτος Ακώστα, το πλήρωσε ο αθλητισμός και μερικοί ε, ασχολούμενοι με το βόλεϊμπολ, οι οποίοι τιμωρήθηκαν και δεν μπορούσαν καν να εισέλθουν στον λέσχη τους, αθλητική του λέσχη. Οι συνέπειες ήταν ε, πολύ σκληρές ο πρώην πρόεδρος του Βέλμπολ τη Αργεντινή, Μόραν Γκόιμαν, άρχισε να επικρίνει τον Ρούμπερ Κώστα όταν, ε, μάλλον στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2002. Και ο Ακώστα αποκλείστηκε από την ε, Ομοσπονδία της Αργεντινή και χρειάστηκε να καταβάλει περίπου 800.000 δολάρια ως ε, πρόστιμο. ο Μάριο Γκόιμεν σήμερα από οικονομικής και ψυχολογικής πλευράς έχει γίνει ράκος. Ε, εξεδιώχθη από την, από την οικία του και δεν μπορεί να ε, πληρώσει τα ιατρικά του έξοδα. Εν τω μεταξύ μεγάλα ποσά σε μισθούς ε, και πριν μετά από τις εκλογές ε, της, στην τι τις πρώτες ε, δημοκρατικές εκλογές μετά από 25 χρόνια. Το handball για 12 χρόνια διοικήθηκε από τον Αιγύπτιο Χασάν Μουσταφά, ο οποίος ε, ταξίδευε για, κατέβαλε έξοδα ταξιδίου πάνω από 400.000 ευρώ χωρίς να ε, υποβάλει κανένα, καμία απόδειξη καν... και είχε παρέμβει σε διάφορες επιχειρήσεις anti-dumping και αντικατέστησε μια σειρά από αξιωματούχους όταν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Handball ο ε, συνεδρίασε ο πρόεδρος Χασάν Μουστάφα φρόντισε να μην ε, πάρουν το λόγο οι συμμετέχοντες και ε, υπερψηφίστηκε και επανεξελέγει με συντριπτική πλειοψηφία. Όλοι γνωρίζουμε το σκάνδαλο ISL. ISL ήταν μια επιχείρηση για την, που εκμεταλλευόταν τα δικαιώματα εκπομπών τηλεοπτικών. Και από το 89 στο 2001 η ISL πλήρωσε τουλάχιστον 160 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα για λαδώματα. Γνωρίζουμε τώρα μερικά από τα πρόσωπα τα οποία έλαβαν χρήματα, δωροδοκήθηκαν από την FIFA. Αλλά να έχετε πει ότι 90% από τα 100 εκατομμύρια ε, χρήματα τα οποία δόθηκαν σε μίζες δεν έχουν ακόμα διερευνηθεί. Ορισμένα από τα πρόσωπα αυτά ακόμα μπορούν να έχουν ε, κάποια υψηλά αξιώματα. Το IOC ξεκίνησε κάποιες μεταρρυθμίσεις το 1999 για να ανταποκριθεί στις ε, εκδηλώσεις αυτές. Ε, υπάρχουν τώρα κάποιοι κανόνες καινούργοι έτσι ώστε κανένα μέλος της IOC μην είναι σε θέση να δωροδοκηθεί. Παρά το ότι ε, μια σειρά από ε, αρχές Επίσης στην περίπτωση της FIFA ε, ασχήθηκε μαζική πίεση για να ξεκινήσει μια διαδικασία μεταρρύθμισης την οποία σίγουρα θα έχετε ακούσει. Τώρα που οδηγούν όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις θα δείτε ότι υπάρχουν ε, αντιφατικές απόψεις, αντιφατικές απόψεις από τις ε, σχολές που υπάρχουν ε, από το 1976 υπήρξε μια σχολή η οποία στήριξε το διεφθαρμένο αυτό σύστημα αλλά και επίσης ε, έχει αποφασιστεί ότι το σύστημα δεν μπορεί να, να τροποποιηθεί χωρίς να μεταρρυθμιστεί η FIFA. Αυτό που είναι σίγουρο είναι αν εσείς και εγώ ε, πάψουμε να, να ελέγχουμε την FIFA δεν θα μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε χρήματα. Τώρα οι συζητήσεις οι οποίε ε, οργανώθηκαν πρόσφατα, οι δύο βασικές μεταρρυθμίσεις ε, της ε, FIFA ζητήθηκε να δοθεί έμφαση τους όρους critical και accompaniment. Όλοι σε αυτό την αίθουσα σίγουρα συμφωνούν πως μια ανεξάρτητη οργάνωση είναι ένα βασικός παράγον στην σημερινή μας εποχή. Θα πρέπει λοιπόν να καταπολεμηθεί η διαφθορά και το έγκλημα από αυτούς οι οποίοι δεν τηρούν κανέναν από τους βασικούς κανόνες της κοινωνίας έφτασε η ώρα λοιπόν για εσά ω πολιτική να αντιδράσετε στα όσα συμβαίνουν στον αθλητισμό. Και τέλο, να αναφερθώ σε κάποιε δράσει που δεν μπορούσατε να αναλάβετε χωρί να επηρεάσετε την αυτονομία του, του αθλητισμού. Είναι δικαίωμά σα και υποχρέωσή σα να προστατέψετε του φορολογούμενου και τα χρήματά του. Τα αθλήματα λαμβάνουν σημαντικές, σημαντικά ποσά, ε, επιδοτήσεις ε, για τις ε, αθλητικές ε, εκδηλώσεις ε, αλλά και για τις διάφορες εγκαταστάσεις. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να φροντίσουν ώστε να υπάρξει και το κατάλληλο πνεύμα στους, στον αθλητισμό. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να διατηρηθεί η πίεση από τις Ευρωπαϊκέ και ε, διεθνεί ε, αθλητικές οργανώσει, ζητώντα από τον ISL μια εξέταση όλων των περιπτώσεων όπου έχουν διαπιστωθεί ε, προσπάθεια επιρροής Κάποιες από αυτές τις δράσεις ε, προωθούνται από την οργάνωση Play the Game στη Δανία και από κάποιες αθλητικές οργανώσεις σε συνεργασία με έξι ευρωπαϊκά πανεπιστήμια συμπεριλαμβανομένων των ε, ε, Αθλητική Ακαδημία της Γερμανίας. Θα παρουσιάσουμε ένα εργαλείο για τον Απρίλιο και θα σας καλέσουμε να παρευρεθείτε σε αυτή την εκδήλωση. Και κάτι άλλο που θα μπορούσε να βελτιώσει το κλίμα είναι να διοργανώσουμε μια ε, διάσκεψη για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Εστάλλη. μάλλον το 2011 υπήρξε μια διάσκεψη στην κολονία, αλλά μέχρι τώρα η IOSC δεν έχει αντιδράσει. Μπορείτε να επιμείνετε επίση για την βέλτιστη διακυβέρνηση στον αθλητισμό τουλάχιστον σε δύο εκδηλώσεις του 2013, την ε, ΜΙΝΕΠΣ 5 που θα εξαρθεί στο Βερολίνο τον Μάιο και το δική μας στη Δανία δηλαδή, ε, Play the Game 13. Τέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, η Ευρώπη θα πρέπει να ηγηθεί στην δημιουργία ενός γραφείου συμψηφισμού, ένα όργανο το οποίο θα παρέχει αλλά και θα είναι χώρο ανταλλαγής πληροφοριών για την καταπολέμηση διαφθοράς στον αθλητισμό κυρίε και κύριοι. Φαίνεται ότι ε, τα λόγια του Τάμας Ατζάν ε, εισακούστηκαν και θα, θα προχωρήσουν προς ε, με ένα αθλητισμό με, χωρίς μάλλον διαφθορά και τη δυνατότητα συνεργασίας. Ευχαριστώ. Thank you very much. It was... Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ε, πολύ απογοητευτικό η κατάσταση που περιγράφατε ακούγοντά σα και πρέπει πράγματι κάτι να κάνουμε. Πρέπει να ξέρετε όμως ότι δεν είμαστε τόσο πανίσχυροι. Η Επιτροπή μας δεν έχει μεγάλη δύναμη. Έχει ωστόσο την υποχρέωση να σας ακούσει και να προσπαθήσει να σας βοηθήσει με τον ΑΒ τρόπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Και παρόλο που υπάρχουν απόντες, ξέρω ότι είναι καλό να τους ακούσουμε μια μέρα. Έχουμε πολλές παρεμβάσεις πριν να δώσω το ε, μικρόφωνο στην αίθουσα θα ήθελα να χαιρετήσω τον κύριο Μαυρομάτη που ήρθε εδώ χαίρομαι που σας βλέπω για να μας μιλήσει λοιπόν Σαντιάκο Πίσερ παρακαλώ Ευχαριστώ Πρόεδρε Έχοντας ακούσει τα όσα μας είπαν οι προσεκλημένοι έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας δεν ξέρω αν θα έχουμε τις αρμοδιότητες για να προχωρήσουμε. Θα ήθελα ε, έχουμε να μιλήσω για πολλά σημεία και μάλλον θα τα μπλέξω. Αλλά σύμφωνα με τα όσα άκουσα, επίσης ότι υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα. Πρώτα απ' όλα, όταν ε, μιλάμε για τα στοιχήματα, θα πρέπει να κάνουμε διαφοροποίηση ανάμεσα στο νόμιμο στοίχημα και στο θέμα του σήματος των παιχνιδιών, που είναι πράγματα διαφορετικά. Αν προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις ε, για τα ζητήματα αυτά στην έκθεση που θα ψηφίσουμε για τον αθλητισμό προκύπτουν κάποιες ιδέες δηλαδή να υπάρξει ένα ε, ευρωπαϊκό αδίκημα για τον αθλητισμό θα πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη να το συμπεριλάβουν στον ποινικό του κώδικα και αυτό θα σημαίνει για, όχι μόνο για τα στοιχήματα αλλά και για την διαφθορά στους διάφορους ε, αθλητικούς οργανισμούς, ενώσεις, ε, συλλόγους, αθλητικούς κλπ. Διότι αυτά έχουν τεράστιες ε, οικονομικές ε, και ηθικές επιπτώσεις. Αν υπάρχει λοιπόν διαφθορά, αυτό έχει επιπτώσεις και στον οικονομία και στον τουρισμό και σε άλλους κλάδους. Ε, αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι ζήτημα πολύ σημαντικό. Μία από τις ιδέες που συμπεριπελαμβάνονται στην έκθεση είναι το ζήτημα της πνευματικής ιδιοκτησίας για διάφορα αθλητικά γεγονότα. Δηλαδή, εάν εγώ οργανώσω ε, ένα πρωτάθλημα, φυσικά ο διοργανητής έχει το δικαίωμα του merchandising. Μπορεί δηλαδή να πουλήσει τα δικαιώματα στις τηλεοράσεις, φυσικά τηρώντας το δίκαιο της, στην πληροφόρηση. Αλλά εμείς έχουμε αυτήν την ε, δυνατότητα σε, όλα τα, σε όλες τις διοργανώσεις που γίνονται. Αλλά θα πρέπει να μπορούμε να ελέγχουμε ποιοι είναι αυτοί που μπορούν να στοιχηματίζουν στα γεγονότα αυτά και ποιοι όχι. Αλλά δεν μπορούν όλες οι οργανώσεις ε, να οργανώνουν ε, στοιχήματα. Υπάρχουν επίσης στοιχήματα αθλητικά τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τον αθλητισμό, η περίπτωση του κρίκετ υπενθυμίζω. Την οποία γνωρίζω πολύ καλά. Υπήρχε στήσιμο των ε, παιχνιδιών επανειλημμένα το, κάτι το οποίο δεν έχει σχέση με τους κανόνες του παιχνιδιού ε, ε, γίνονται στοιχήματα εντός ε, ενός ε, αθλητικού γεγονότος. Αν μπορούν λοιπόν να ληφθούν μέτρα για τις περιπτώσεις αυτές. Ο κύριος Μίταγ ε, μίλησε για την οικονομική πτυχή. Θα ήταν πολύ καλό να υπάρχουν κάποια ανώτατα όρια στα γραφεία στοιχημάτων. Εμένα μου αρέσει η όπερα και έχει υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στα μεγάλα ε, θέμα θεατρικές εκδηλώσεις για τα εισιτήρια, να μην μπορούν να λένε υπερβαίνουν τα εισιτήρια πάνω το ένα μια συγκεκριμένη αξία. Στην έκθεση υπήρξε μια τροπολογία ενός συναδέλφου φιλελευθέρου που έλεγε ότι θα πρέπει να περιορίσουμε τον αριθμό των παικτών στις ομάδες έτσι θα περιοριστούν το σύνολο των εξόδων, των δαπανών. Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό ή όχι, αλλά ε, δεν θα είμαστε εμεί αυτοί που θα αποφασίσουν πόσοι παίκτες, πόσοι έχει μια ομάδα. Αυτό εξαρθεί από, την, από τις και από τους κανόνες. για το θέμα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων στην, Ισπανία, τα δικαιώματα αυτά τα έχουν οι αθλητικές λέσχες. Ένα άλλο ζήτημα αφορά τις ε, αθλητικές υποδομές. Εάν ένας Δήμος πληρώσει για την κατασκευή ενός ε, γηπέδου ποδοσφαίρου και το διαθέτει δωρεάν σε μια ομάδα, ε, πρέπει να καταλάβουμε ότι η ομάδα έχει πληρώσει πολλά για να κατασκευάσει αυτό το κτίριο. Ίσως θα πρέπει το γήπεδο. Θα πρέπει και αυτό να δούμε πώς μπορούμε να καλύπτονται αυτά τα έξοδα. Εμείς ε, οργανώνουμε τα εμπορική αν θέλετε εκδήλωση στο πλαίσιο ε, μιας αθλητικής διοργάνωσης ε, σε στυλ ε, NBA της Αμερικής και να πω ότι οι διάφορες λέγγες που υπάρχουν στην Ευρώπη θα μπορούσαν να συνεργαστούν, αυτό θα πρέπει να μας, ε, μάλλον θα πρέπει να μας οδηγήσει στο να ε, ρυθμίσουμε και τα θέματα τα οικονομικά. Τώρα, ε, να καταλήξω ότι το θέμα της διαφθοράς δεν αφορά μόνο τα στοιχήματα, αλλά και τις αποφάσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο των, των αθλητικών συλλόγων. Εγώ συζήτησα με τον κύριο Μπλάτερ και μου επέστησε την προσοχή γιατί όταν οργανώνουν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Τέλος, αν υπάρξει κάποια ομάδα, κάποια λέσχη που δεν διαφωνεί με μια απόφαση, τότε χρειάζεται, θα πρέπει να υπογράψει μια ε, σύμβαση για, συμμετω... την συμμετοχή της σε αυτήν την ε, διοργάνωση. Υπάρχει τώρα ε, η δικαιοσύνη, η αθλητική, αλλά και η τακτική δικαιοσύνη. Ε, εγώ, ήθελα να συσταθεί ένα ευρωπαϊκό δικαστήριο στο Λουξεμβούργο π.χ. για να εξετάζει τις διάφορες ε, περιπτώσεις και το δικαστήριο αυτό να είναι στην Ευρώπη, να μην είναι στην ε, Ελβετία όλες οι οργανώσεις, όλα τα, όλοι οι σύλλογοι ε, δέχτηκαν κάποιες απειλές και θεώρησαν ότι δεν είναι ορθές πάντα οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το δικαστήριο της Ελβετίας. Γι' αυτό λοιπόν εκείνη την πρόταση που είχα κάνει για το ελευθερικό Δικαστήριο την απέσυρα από την έκθεση που είχα συντάξει. Τώρα φυσικά οι συνάδελφοι που θα ακολουθήσουν θα μπορούν να περισσότερο κάποια σημεία. Ευχαριστώ Ιβο Μπέλετ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Πρόεδρε, χωρίς μικρόφωνο ο κύριος Μπέλετ. δυο τρει ερωτήσει. Πρώτα απ' όλα στον κύριο Γκάρλικ. Πράγματι, όπως είπατε κύριε Πακ, είναι ανησυχητικά αυτά τα οποία ακούμε. Είναι μεγάλος κίνδυνος για το μέλλον του επαγγελματικού αθλητισμού. Αλλά θέλουμε να ακούσουμε περισσότερο το τι μπορεί να κάνει η Europol. Πώς μπορεί να βοηθήσει και πώς μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε. Αναφερθήκατε το ότι οι περισσότερε περιπτώσεις, ε, οι περισσότεροι αγώνες στείνονται στην Ασία. Μήπω είμαι χαμένη υπόθεση από την αρχή. Και επίση ε, η Europol ε, ανταλα... λαμβάνει τα δεδομένα που ανταλλάσσουν τα 27 κρατημέλη. Υπήρχε ειδικά τα συστήματα έγκαιρη προειδοποίηση που έχει φτιάξει ο τομέα. Είστε κι εσεί μέσα σε αυτό το σύστημα. Ήδη κάποιες πρωτοβουλίες λαμβάνονται στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Κομισιόν είναι εδώ, το Συμβούλιο. Τι πρωτοβουλίες μπορούν να αναλυφθούν για να βοηθήσουμε ένα τον άλλον για να αντιμετωπίσουμε αυτό τον σοβαρό κίνδυνο για τον επαγγελματικό αθλητισμό. Δεύτερον, κύριε Γκάλεκ, μιλήσατε για τους μάνατζερ των παιχτών, γιατί η Κομισιόν έκανε πριν από δύο χρόνια μία μελέτη για το θέμα αυτό και ε, εκεί υπήρχαν κάποια ανησυχητικά στοιχεία. Μπορείτε να μας πείτε κάποια πράγματα. Η Europol ε, έρευνα και ύποπτες ε, χρηματικές ροές όσον αφορά τους μάνατζερ των παιχτών. Ο κύριος μάνατζερ, ο κύριος Άντερσον αναφέρθηκε στην FIFA. Μπορείτε κύριε Γκάρλικ να μας πείτε κάτι περισσότερο για την έρευνα της FIFA και μπορεί η Europol να παίξει ένα πιο προληπτικό ρόλο σε σχέση με την πιθανή απάτη εντός της FIFA. Και τέλος, αν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, έχω άλλες δύο ερωτήσεις προς τον κύριο Δόκτωρα Μίταγκ. Συμφωνώ μαζί σας πως το Financial Fair Play είναι πολύ σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, όμως αναφερθήκατε στην περίπτωση της Manchester City και στην χορηγία των 400 εκατομμυρίων ευρώ, ε, που σημαίνει πως ε, ήδη το σύστημα αυτό παρακάμπτεται με τρόπο πολύ δημιουργικό. Οπότε τι θα κάνουμε. Και ο κ. Φίσας επίσης αναφέρθηκε στα δικαιώματα τα τηλεοπτικά, που είναι μεγάλο στοιχείο δεν θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη αλληλεγγύη εντός του ποδοσφαίρου με την ενίσχυση της οικονομικής αλληλεγγύης στο Champions League. Ήδη υπάρχει οικονομική αλληλεγγύη, αλλά οι μεγάλες ομάδες των μεγάλων πρωταθλημάτων που είναι εκεί πέρα τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δικαιώματα λαμβάνουν πολύ περισσότερα από τις άλλες. Χρειάζεται μεγαλύτερη αναδιανομή των ε, εσόδων ε, των τηλεοπτικών. Και τέλος, κυρία Πρόεδρε, ο Σαντιάγκο το ανέφερε, πιθανό πλαφόν στο ποσό των μεταγραφών. Ή ίσως μια άλλη ιδέα, περισσότερη αλληλεγγύη όσον αφορά τα έσοδα των μεταγραφών. Ε, σε ένα κοινό σύστημα. περισσότερη αλληλεγγύη στις μεταγραφές. μπορείτε ίσως να κάνετε κάποιες προτάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Πέτρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει η κυρία Καμερέβερτ. Για αυτά τα οποία μας είπατε. Είχαμε διαβάσει κάποια από αυτά στις ε, εφημερίδες ε, και έμοιαζαν με αστυνομικό μυθιστόρημα. Αλλά θέλω να ξεκινήσω με τον κύριο Γκάλε. Είπατε πως ε, πολλοί αγώνες στείνονται ε, εκτός Ευρώπης, κατά βάση στην Ασία. Αλλά βεβαίω οι επιδράσεις μετά είναι εδώ στην Ευρώπη. Οπότε το ερώτημά μου είναι πόσο καλή είναι η συνεργασία ε, των διεθνών αρχών με την ε, Europol ε, και με τις εθνικές αρχές ε, αλλά και με την Interpol στην Ασία ή οπουδήποτε αλλού. Το άλλο ερώτημα. είναι πως υπάρχει και διαφθορά εντός των ομάδων. Οπότε το ερώτημα είναι έχουν οι ερευνητικές αρχές την δυνατότητα να παρέμβουν ή είναι ε, ζήτημα αυτορύθμισης ε, των ομοσπονδιών. Αν τα αφήσουμε στις ομοσπονδίες, το επόμενο ερώτημα είναι ποιες ε, δυνατότητες βλέπετε νομοθετικές για παρέμβαση με τις περιορισμένες δυνατότητες που έχουμε εμείς με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας. Μπορούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσουμε ως Κοινοβούλιο. Το επόμενο ερώτημα αναφέρεται στο Financial Fair Play. Και εγώ θεωρώ πως είναι βήμα σε σωστή κατεύθυνση αυτό το οποίο έχει κάνει η UEFA. Αλλά ακούγοντας αυτά τα οποία είπατε, κύριε Μίταγκ, διαπιστώνουμε πως ε, υπάρχουν ε, ήδη ε, κάποια παραθυράκια και δεν επαρκεί το σύστημα. Π.χ. είπατε υπάρχουν 6.000 επαγγελματικέ ομάδες που έχουν κάποιο είδου άδεια στην Ευρώπη. Αλλά στο Financial Fair Play βεβαίω υπάγονται οι ομάδες οι οποίες παίζουν στην Ευρώπη μόνο. Οπότε μειώνεται αυτομάτως ε, ο αριθμός αυτών που πρέπει να ενταχθούν σε αυτούς τους ε, κανόνες. Δηλαδή μιλάμε πόσο για καμιά κατοσταριά ομάδες. Ποιες ε, δυνατότητες βλέπετε για να επεκταθεί αυτό το σύστημα. Και αναφέρατε και άλλα προβλήματα. Ε, φαίνεται πως ε, πρόοδος εδώ πέρα είναι πάρα πολύ αργή, ειδικά αν δούμε τις μεταβατικές ε, περιόδους που υπάρχουν στο Financial Fair Play. Δηλαδή και οι ρυθμίσεις που έχουμε τώρα δεν ξέρω κατά πόσον θα είναι αποτελεσματικές. Αναφέρατε και εσείς ήδη τα, τα παραθυράκια. Βλέπετε ανάγκη, δυνατότητα από τη δική μας την πλευρά, την πολιτική την πλευρά, είτε σε ευρωπαϊκό είτε σε εθνικό επίπεδο να στηρίξουμε αυτή τη δικασία και να προωθηθεί λίγο. Δεν ξέρω αν έχουμε καν τέτοια δυνατότητα, αλλά θα ήθελα τη δική σας την εκτίμηση για το τι μπορούμε να κάνουμε. Να απευθύνουμε η έκκληση και στην ΟΕΦΑ και σε άλλες ομοσπονδίες Βλέπετε κάποια δυνατότητα, λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε. Και όπως είπα και νομοθετικά να το πλησιώσουμε. Ευχαριστώ, Μάρτιν Λόκερκάρτ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριοι, για τις αναλυτικές και πιστικές παρουσιάσεις σας. Όποτε σας ακούω, φαίνεται πως συσσωρεύονται και άλλα πράγματα πέρα από αυτά που ξέρουμε και είναι ανησυχητικά. Οι συνάδελφοι είπαν ήδη κάποια πράγματα και πρέπει να συμφωνήσω. Πρώτον, ένα ζήτημα που αναφέρατε και ο κύριος Γκάρλικ το είπε, είπατε πως οι συνάδελφοι δηλαδή ρώτησαν εάν έχετε καμία συνεργασία με τις τοπικές αρχές στην Ασία. Όλοι ξέρουμε πως είναι σημαντική η διαφθορά στην ε, Κίνα και δεν ξέρω αν έχετε κάποιες επαφές εκεί για να κάνετε κάτι. Ε, αν ισχύει κάτι τέτοιο δεν ξέρω. Μετά είχαμε την παρατήρηση για τα βορειοευρωπαϊκά πρωταθλήματα έχετε την εντύπωση πως ε, ε, ε, υπάρχει μια έρευνα εκεί πέρα σε τοπικό επίπεδο. Επίσης, κατά την άποψη σας, ποιο είναι σήμερα το μεγαλύτερο εμπόδιο στη δουλειά σας. Θα ήθελα και αυτό να το μάθω. Γιατί φαίνεται πως κάνετε πολλά, αλλά βεβαίως αντιμετωπίζετε και προβλήματα. την ανησυχία σας για τις ε, εθνείς αθλητικούς οργανισμούς. Και γιατί για μας είναι ακόμη πιο δύσκολο να μιλήσουμε, γιατί όταν τους μιλάμε βλέπω πως δεν ε, έχουν και πολύ όρεξη. Να αν την ίδια αντιμετώπιση βλέπετε κι εσείς. Έχετε ιδέα αν αυτό σχετίζεται και με το πολιτικό επίπεδο. Θα ήθελα να ακούσω και τα σχολιά σας γι' αυτό. Και τέλος, προς τον κύριο Άντερσεν. Πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Δύο προτάσεις ε, έχετε. Η μία ιδιαίτερα τράβηξε ενδιαφέρον. Ε, αυτό το οποίο αναφέρατε κάπου να γίνεται μια κεντρική εκαθάριση. Ίσως ε, αυτό θα μπορούσε να μας ε, βοηθήσει. Είναι ενδιαφέρουσα ιδέα. Αν μπορούσατε λίγο να επεκταθείτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Μπουσκούρτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι έχουμε τόσο επιφανείς προσκεκλημένους που μίλησαν τόσο ειλικρινά για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Uh, um, uh, για την ακαιρεότητα στον αθλητισμό είχαμε πέρσι και την έκθεση φύσας ε, στην Επιτροπή Ελευθεριών. Είχα γράψει τη γνωμοδότηση εγώ, ειδικά αυτή την πτυχή δηλαδή της απάτης στον αθλητισμό και ένα από αυτά τα οποία είπα ε, ήταν το ότι εσωτερικά και εξωτερικά πρέπει να υπάρχει μηδενική ανοχή στη διαφθορά. Γιατί η διαφθορά δεν είναι μόνο εξωτερική αλλά και εσωτερική εντό των ομοσπονδιών. Οι νομοσπονδίε ε, και οι οργανισμοί του ποδοσφαίρου δεν είναι πάνω από τον νόμο. Τι μπορεί να, συγκεκριμένα τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε εμεί, όπω ρώτησαν και οι συνάδελφοι, ειδικά όταν μιλάμε για τις ε, ομοσπονδίες που δίνουν κάποιες άδειες ε, σε υπεργολάβους ε, πώς μπορούν να ελεγχθούν ε, καλύτερα. Ποιοι είναι οι έλεγχοι όσον αφορά την ακαιρεότητα. Βεβαίως όλοι ξέρουμε την κατάσταση στη FIFA με την διεθνή διαφάνεια που κάποια στιγμή είπε πως εντάξει φτάνει τα παρατάμε. Νομίζω πως είναι σημαντικό να δούμε το μέλλον του αθλητισμού. Η ακαιρεότητα να αποτελέσει βασικό ζήτημα πριν καταστραφεί το άθλημα. Βεβαίω είναι και ζήτημα νομικό, έτσι, όχι μόνο αθλητισμού. Οπότε, αυτό το οποίο θα ήθελα να ρωτήσω είναι πώς μπορούμε εμείς να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Όχι μόνο η Υπουργοί Αθλητισμού και οι οργανώσεις ε, και οι οργανισμοί του αθλητισμού, αλλά και η δικαιοσύνη, η αστυνομία. Και αυτό το οποίο λείπει νομίζω είναι ο συντονισμός, παραδείγματος χάρη στο στήσιμο των αγώνων. Ε, είχα γράψει και μία έκθεση τον προηγούμενο μήνα για την Επιτροπή Οργανωμένου Εγκλήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και αυτό το οποίο είπα είναι πως γίνονται ήδη κάποια πράγματα με του ενδιαφερομένου, με του οργανισμούς του αθλητισμού, αλλά που είναι ο συντονισμός. Γιατί ναι, είναι παγκόσμιο πρόβλημα, είναι όνειρο να σκεφτόμαστε πώ θα το λύσουμε, αλλά στο ευρωπαϊκό επίπεδο κάτι μπορούμε να κάνουμε. Και υπάρχει βεβαίως και η δουλειά του Συμβουλίου της Ευρώπης για το στήσιμο των αγώνων, αλλά νομίζω πως και η Ευρωπαϊκή Ένωση η ίδια που έχει περισσότερα μέσα ε, μπορεί να νομοθετήσει κτλ. Ε, πρέπει να κάνει περισσότερα. Θέλω να ακούσω και τις δικές σας τις σκέψεις. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τις δικές σας σκέψεις για μια λύση. Γιατί πρέπει να συντονιστούμε. Uh, Ευχαριστώ. Εμινέ. Μπόρις. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την παρουσίαση. Ε, Τα ζητήματα που θίξατε είναι νομίζω ζητήματα που μας ενδιαφέρουν και φυσικά ενδιαφέρουν και άτομα τα οποία εμπλέκονται σε τα, στα αδικήματα αυτά. Υπάρχει άρθρο στη συνθήκη που μας δίνει την θεωρητική δυνατότητα τουλάχιστον να αντιμετωπίσουμε και να καταπολεμήσουμε κάποιες ε, από αυτές τις αντασταλίες. Φυσικά για τους νομομαθείς, για όλους μας ε, είναι απαραίτητη μια ανάλυση, μια εξέταση αυτού του παθολογικού ζητήματος ε, της παθολογίας ε, και πώς θα μπορούσε να διευθετηθεί και να ρυθμιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιστεύω ότι σήμερα πλέον ο αθλητισμός έχει διεθνοποιηθεί και είναι δύσκολο να περιοριστούμε μόνο σε, στις ευρωπαϊκές αρμοδιότητες, διότι παραδείγματος χάρη η UEFA ε, περιλαμβάνει μια σειρά από ευρωπαϊκές αλλά και μη ευρωπαϊκές ε, οργανώσεις Χρειάζεται όμως εμείς να εμπνεύσουμε κάποια δράση. Γι' αυτό απαιτείται μια διεθνής ε, συνδιάσκεψη όπως συμβαίνει για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, πρωτόκολλο του Κιώτο κλπ. Υπάρχει δυνατότητα λοιπόν να προωθήσουμε μια πραγματικό προβληματισμό για τον αθλητισμό που έχει επιπτώσεις και σε άλλους κλάδους. για να κοιτάξουμε στον τομέα του ποδοσφαίρου, παρατηρούμε ότι ως επιτοπλίστων επικεντρώνεται το θέμα αυτό στην Ευρώπη. Οι, διάφοροι αγώνες οργανώνονται στην ευρωπαϊκό έδαφος και τα χρήματα που δαπανώνται στον τομέα του ποδοσφαίρου είναι χρήματα ευρωπαϊκά. Ξέρουμε ότι υπάρχει ε, ε, ένα, ένα σύνολο δραστηριοτήτων που εμπλέκονται όπως ε, οι πωλήσει των αθλητικών στολών. Με βάση λοιπόν το άρθρο 165 θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα, τα αρρωστημένα θα μπορούσα να πω, χρειάζεται να οργανωθεί μια παγκόσμια διάσκεψη στην οποία συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Αναφέρθηκε ήδη, είναι απαραίτητο να προωθηθεί κάτι τέτοιο τόσο Μάλλον και θα ήθελα τώρα να επικεντρωθώ σε κάποια στοιχεία όπως η χρηματοδότηση ή καλύτερα το fair play, το οικονομικό εφαγωνίζεστε. Μπορούμε λοιπόν να συνεργαστούμε με την FIFA για να οδηγηθούμε σε μια ρύθμιση των προβλημάτων αυτών που φυσικά η UEFA είναι αυτή η οποία ασχολείται με το οικονομικό εφα, αγωνίζεστε. Αλλά ε, υπάρχουν και ακολουθούνται κάποιοι εθνικοί κανόνες Συχνά πρόκειται για οργανώσεις, για ενώσεις. Κάθε χώρα λοιπόν έχει ένα διαφορετικό σύστημα μέσω του οποίου μπορεί να ελέγχει τους ε, ισολογισμούς των ε, ομάδων ε, αλλά και να εξετάσουν και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται από τις διάφορες αθλητικές λέσχες. απαιτείται ένας κανονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις ε, εμπορικές ε, οργανώσεις ε, κάτι το οποίο θα μας επιτρέπει θα μας επιτρέψει να κάνουμε και τις απαραίτητες συγκρίσεις τώρα για τα τηλεοπτικά δικαιώματα και εδώ πρέπει να είμαστε πιο συνεπείς αλλά και να δείξουμε μεγαλύτερη αλληλεγγύη διότι οι εκπομπές ε, αφορούν τις μεγαλύτερες ε, ομάδες ε, οι οποίες έχουν και τις μεγαλύτερες τις Αργά ή γρήγορα λοιπόν αυτό το ζήτημα θα πρέπει να ρυθμιστεί. Ένα άλλο ζήτημα, η αυτορύθμιση και των μεταγραφών. Δεν είμαι πεπισμένος ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποιο ανώτατο όριο στις μεταγραφές. Δύσκολο μπορούμε να φορεστούμε κάτι τέτοιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα μεγάλο κομμάτι της διαφθοράς γίνεται ακριβώς εδώ. Ε, πάρα πολλά είναι τα σκάνδαλα στα οποία εμπλέκονται ποδοσφαιριστές ε, οι οποίοι μοιράζονται τα χρήματα με όσους είχαν ε, προσπαθήσει να προαγαγούν να προάγουν κάποιε εξελίξεις. Πρέπει να θέσουμε λοιπόν κάποια ανώτατα όρια. Τώρα, αυτό το οποίο ανέφερε ο Σαντιάγκο. Η Πολωνία είναι ένα καλό παράδειγμα σε ό,τι φορά την μεταφορά των οδηγίων. Ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα διαφθοράς στο ποδόσφαιρο την τελευταία 20 ετία. Πραγματικά έγινε στην Πολωνία, στην πατρίδα μου. Και γνωρίσαμε τεράστια, πάνω πολύ υψηλά επίπεδα διαφθοράς. Ε, πολλά άτομα καταδικάστηκαν το 2005 υπήρξαν ε, πρόσωπα τα οποία κατέληξαν στην φυλακή. Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα γενικευμένο θα έλεγα, δεν αφορά μόνο στο ποδόσφαιρο. Τώρα πια το ποτάθλημα στην ε, χώρα μου έχει γίνει ένα πιο διαφανή. Εντάξει, πέρασε από χίλια κύματα, αλλά τώρα τα πράγματα ξεκαθάρισαν. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο τώρα μπορούμε να ενεργήσουμε, μπορούμε να δράσουμε και η Κομισιόν θα πρέπει τουλάχιστον να ε, δώσει έναν ενιο ορισμό. Λοιπόν, έχουμε την υποχρέωση να αντιμετωπίσουμε και να καταπολύσουμε την διαφθορά στον αθλητισμό και να μην υπάρχουν πλέον κατά το δυνατόν στημένα παιχνίδια και στημένα στοιχήματα. Απαιτείται λοιπόν ένας ενίος ορισμός μικρά βήματα τα οποία όμως μπορούν να έχουν σημαντικές συνέπειες. Απαιτείται να στηρίξουμε την, ε, μια, νέα, μια διάσκεψη αλλά και διερωτώ με αν αυτό μπορεί στην πράξη να υλοποιηθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δύο, τρία πραγματάκια να πω κι εγώ. Δεν θεωρώ πως είναι τόσο απλό να πούμε πως εμείς πρέπει να κάνουμε κάτι. Ποιοι είμαστε εμείς καταρχήν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί. Άρα μπορούμε να απευθύνουμε έκκληση στους υπεύθυνου να το κάνουν. Η UEFA προσπάθησε, προσπαθεί, αλλά ξέρετε, λάθη υπάρχουν ε, και τα είπατε κύριε Μίταγκ παντού υπάρχουν παραθυράκια, δεν είναι δυνατή η σωστή παρακολούθηση, ε, αλλιώς θα είχαμε ένα τεράστιο μηχανισμό. Οπότε δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, αλλά καλό είναι να το συζητήσουμε. Το ερώτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να ενημερώσουμε εμείς κάθε μέρα, να ευαισθητοποιήσουμε διαβάζει κανείς την εφημερίδα, όχι μόνο τη γερμανική και σε άλλε χώρε διαβάζουμε κάθε μέρα, κάθε μέρα για διαφθορά τα μάνατζερ ε, επιχειρηματιών, πολιτικών. Δεν τα συζητάμε αυτά κάθε μέρα. Αυτά τα οποία είπατε εσείς έγινε μία φορά μία μεγάλη ιστορία και μετά εξαφανίστηκε. Μα αυτά έπρεπε να είναι ψωμοτήρι καθημερινά να μας απασχολούν. Βεβαίω ε, θα μπορούσε να υπάρξει μια διεθνή ε, διάσκεψη, αλλά το ζήτημα είναι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Αναφέρατε τη μεγάλη διάσκεψη της UNESCO στο Βερολίνο. Καλό θα ήταν ε, πράγματι κάποιος με ένα σημαντικό όνομα ή μια σημαντική θέση να σηκωθεί και να πει θέλω να αναφερθώ σε αυτό το ζήτημα. και πρέπει να κάνουμε κάτι. Αλλά όπως είπα, εμείς έχουμε περιορισμένες αρμοδιότητες. Αλλά το, να μιλήσουμε μπορούμε να το κάνουμε νομίζω. Και οπωσδήποτε νομίζω μπορεί να, να βγει και στα μήμια. Έχω άλλη μια ερώτηση στους κυρίους της Europol. Ίσως δεν σας κατάλαβα. Είπατε δεν θέμε μηδενική ανοχή ή δεν κατάλαβα καλά. Αυτές ήταν οι παρατηρήσεις μου. Θα δώσω τώρα το λόγο στους ειδικούς. Αλλά δεν θέλω να απαντήσετε όλες τις ερωτήσεις, αυτές οι οποίες αφορούν τον καθένα από εσά. Ποιος θα ξεκινήσει λοιπόν. Europol. Okay. Europol. Μάλιστα, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις. Προσπάθησα να τις σημειώσω. Δεν μπορώ να σας υποσχεθώ πως θα είμαι πλήρως επιτυχής, θα καταβάλω προσπάθεια. Ο ρόλος της Europol είναι να στηρίξει τα κράτη-μέλη. Ε, καταπολέμηση οργανωμένου εγκλήματος και οπωσδήποτε το στήσιμο των αγώνων είναι οργανωμένο έγκλημα. Και βεβαίω ε, στηρίζουμε αυτές τις έρευνες ε, και θα τα συνεχίσουμε αν το ζητήσουν τα κράτη-μέλη. Τώρα, όσον αφορά μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα ειδικών για το ζήτημα, ναι, είναι μια καλή πρόταση. Τα κράτη-μέλη να ορίσουν ικανούς ειδικού που θα μπορούν να πάνε σε συναντήσεις και να, να πηγαίνουν στις συναντήσεις, να ανταλλάσσουν πληροφορίες, βέλτιστες πρακτικές. Θετικό θα ήταν αυτό. Η Interpol ήδη έχει μια παγκόσμια ομάδα εργασία για το στήσιμο αγώνων, στην οποία εκπροσωπείται η Europol. Έχω πάει και εγώ κάποιες φορές ε, στη Λιόν. Ένα από τα ζητήματα νομίζω αφορούσε τις εταιρείε στοιχημάτων και τα δικαιώματα. Δεν είναι η αρμοδιότητά μου. Εμεί είμαστε περισσότερο στην καταπολέμηση του εγκλήματος. Από την εμπειρία μας ξέρουμε πως υπάρχουν πολλά site παράνομα για στοίχημα. Οπότε οτιδήποτε, οτιδήποτε προσπάθεια γίνει για περιορισμό του στοιχήματος πιθανώς θα έχει αποτέλεσμα, αλλά θα οδηγήσει τον κόσμο στα παράνομα site, από τα οποία υπάρχουν χιλιάδες, ειδικά στην Ασία. Αυτή τη στιγμή η Europol στηρίζει μια κοινή ερευνητική ομάδα και θα εξετάσουμε οι μελλοντικέ προτάσεις ε, ε, για επιχειρήσεις. Ε, βεβαίως δεν μπορώ να δεσμευτώ γιατί εξαρτάται και από τους σπόρους. Ε, αλλά τους τελευταίους 18 μήνες κάτι κάνουμε. Και θεωρώ πως είχαμε κάποια επιτυχία στην επίτευξη των στόχων και ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε. Όσον αφορά τις σχέσεις με την Ασία, η Europol προφανώς δεν έχει συγκεκριμένες συμφωνίες που διευκολύνουν την ανταλλαγή ε, στρατηγικών ή επιχειρησιακών πληροφοριών με ασιατικές χώρες. Οπότε από τη δική μας σκοπιά είναι δύσκολο να αντιμετωπίσουμε και να έρθουμε σε επαφή με ε, ασιατικές χώρες άμεσα. Βεβαίως μπορούμε να έρθουμε σε επαφή μαζί τους μέσω της Interpol και οι χώρες που είναι μέλη της Europol μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους διάβλους ε, για τις έρευνές τους και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το δίκτυο συνδέσμων που υπάρχει, που έχουν κάποιες χώρες σε χώρες της Ασίας. Ένα από τα ερωτήματα αφορούσε τους μάνατζερ των παιχτών. Αυτό οπωσδήποτε είναι κάτι το οποίο συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα. Φαίνεται πως κάποιοι ε, μάνατζερ έτσι ακολουθούνται από μια οσμή ε, στισίματος αγώνων ε, και κάποιοι παίκτες ειδικά σε όποιο πρωτάθλημα και αν πάνε. Οπότε, ναι, είναι ενδιαφέροντες οι μάνατζερ, αλλά για πολλά ζητήματα, όχι μόνο για το στήσιμο των αγώνων. Ένα άλλο ζήτημα αφορούσε την ε, FIFA και διαφθορά εντός της FIFA. Όπως είπα, εμείς ασχολούμαστε με το οργανωμένο έγκλημα ε, στα κράτη-μέλη. Οπότε δεν νομίζω να έχουμε την αρμοδιότητα να ερευνήσουμε τη FIFA. Αν το έκανε ένα κράτος μέλος βεβαίως, ε, οπωσδήποτε θα του υποστηρίζαμε με το να δώσουμε ανάλυση και επιχειρησιακή στήριξη και μια πλατφόρμα βέβαια για ανταλλαγή πληροφοριών. Αλλά όσον αφορά την δική, να ξεκινήσουμε δική μας έρευνα είναι απίθανο. Δεν νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο. Η συνεργασία τώρα. Πάρα πολύ καλή. Έχουμε τακτικές συναντήσεις και με την Interpol και χρησιμοποιούμε, όπως είπα, τους διάβλους Τη Ίντερπολ για την Ασία και δεν υπάρχει νομική βάση αυτή τη στιγμή για συνεργασία για στρατηγικά και επιχειρησιακά ζητήματα. Το επόμενο ζήτημα. Ποια είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια. Δεν ανέφερα πως επίσης δεν ανέφερα τις ομοσπονδίες των αθλημάτων ε, γιατί δεν θέλουν να ασχοληθούν με το ζήτημα. Οπωσδήποτε η FIFA έχει δώσει πολλά λεφτά για να ξεκινήσει η Interpol να καταπολεμά το ζήτημα. Οπότε τα στοιχεία λένε πως ανησυχούν. Γιατί ε, σαφώς ε, διακυβεύονται και μεγάλα εμπορικά συμφέροντα αν εμείς διαπιστώσουμε πως υπάρχει τεράστιο ζήτημα διαφθοράς, ε, τότε ο εμπορικός αντίκτυπος θα ήταν ε, τεράστιος. Και θα είχε αρνητικό αποτέλεσμα στο, στο άθλημα που όλοι αγαπάμε. Δεν, δεν λέω ότι είναι έτσι όλοι τόσο διεφθαρμένοι όσο ακούγεται, αλλά κάποιοι είναι. Κάτι άλλο. Τώρα για την Δανία και για τα πρωταθλήματα της Βορείου Ευρώπης. Προσφάτως έγινε μια μεγάλη έρευνα που είχε απήχηση και στον τύπο και σε ανοιχτές πηγές. και αφορούσε στήσιμο αγώνων στο Ροβανιέμι, στη Βόρεια Φιλανδία και οδήγησε συλλήψεις παιχτών και προπονητών και του ανθρώπου που έστησε τον αγώνα. Οπότε ήταν μεγάλη έρευνα. Και έχω δει και κάποια δραστηριότητα στην, στην Νορβηγία. Και το είπα και πριν στην παρέμβασή μου για το σκανδιναβικό ποδόσφαιρο, τα σκανδιναβικά πρωταθλήματα, ότι είναι ελκυστικά γιατί παίζουν μπάλα το καλοκαίρι εκεί πέρα και, ε, και, και οι αμοιβέ είναι επίσης χαμηλότερες. Πώς να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί και να συνεχίσουμε τις έρευνες μας. Νομίζω ότι κάπως βελτιώνουμε την κατάσταση προσπαθώντας, όπως το ανάφερα και προηγουμένως, ε, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα και έχοντας τη σωστή συνεργασία, το μεγάλο ποσό συνεργασίας μέσα στην Ευρώπη, μέσα στα κράτη-μέλη που έχουν το πρόβλημα, νομίζω ότι δεν θα ήθελα, θα δίσταζα να πω ότι υπάρχουν εντελώς αναποτελεσματικά κράτη-μέλη. Δεν υπάρχουν πάνω σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα. Η εμπειρία μας δείχνει ότι πραγματικά είναι καθολικό έγκλημα, καθολικό οργανωμένο έγκλημα και πρέπει να γίνουμε και γινόμαστε αποτελεσματικοί ως σημείο. Το θέμα του συντονισμού των ερευνών είναι πολύ σημαντικό. Έχει αναλυφθεί σε επίπεδο Ευρωπόλ, αλλά υπάρχει ένα θέμα υποστήριξης από τα κράτη και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το προωθήσουμε. Και μετά πολλά πράγματα έχουν αναφερθεί για την πολύ καλή ιδέα των εμπειρογνωμόνων οι οποίοι έχουν ε, ε, την επιθυμία να συγγράψουν ένα εγχειρίδιο για τις ε, χριστότερες πρακτικές για αυτή την καταπολέμηση της διαφθοράς Καταλαβαίνω ότι είχαν δώσει διάφορα παραδείγματα για την Πολωνία και για, ε, για την παρουσίασή τους. Ο Πολωνός ερευνητής είχε ε, καταθέσει μια μαρτυρία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ε, και που μας διαφώτισε ιδιαίτερα. Τελικά πρέπει να πούμε ότι σε σχέση με το επίπεδο ανοχής ε, εγώ είμαι κατά, εντελώς κατά. Μάλιστα μπορώ να πω ότι υπάρχουν σε όλες τις ομάδες καινούργοι παίκτες οι οποίοι επιλέγονται από τους αρχαιότερους παίκτες και η κατάσταση βεβαίως έχει ως εξής. Αν ακούσουν, εγώ πήρα λεφτά για να κάνω το εξής, για να δράσω κατά αυτόν τον τρόπο κτλ. Δημιουργεί ένα είδος καριέρας το οποίο τους ε, είναι ήδη έτοιμο. Και κάποιος ε, ο οποίος έχει δει τα τελευταία χρόνια να τεκταίνονται διάφορα μέσα στα, στους αγώνες και στα παιχνίδια, να εστίσνονται οι αγώνες, είδε πάρα πολλά στισίματα αγώνων μέσα στα χρόνια, τότε ε, ε, μπορεί να ε, ε με αυτή την εμπειρία να ε, παρέμβει και πολύ πρόσφατα είχαμε ένα διάλογο μεταξύ παλαιών και νέων παικτών για το bowling και είπε σε κάποιος αρχαιότερος συνάδελφος έναν νεότερο θα έπρεπε να ξέρεις καλύτερα τι συμβαίνει. Οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να μπορούν να μιλάνε, θα πρέπει να μπορούν να δίνουν τις πληροφορίες που έχουν. Ε, για να είναι δυνατόν να καταλάβουμε πώς λειτουργεί το δίκτυο. Η παροχή της πληροφορίας είναι πολύ σημαντική γιατί είναι ένα θετικό στοιχείο που μας επιτρέπει να προωθήσουμε όλα μας τα θέματα και να φτάσουμε κάπου. Δεν μπόρεσα να σας τα αναφέρω όλα όσα ξέρω, μπορεί να είχα και παραλήψεις και βεβαίως θα απαντήσω σε ερωτήσεις πολύ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριο Σμίταγκ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά το financial fair play είδαμε δύο πτυχές, το ένα βεβαίως αφορά την αλληλεγγύη, το άλλο τις συστάσεις. Νομίζω πως μπορώ να είμαι σχετικά σαφής. Το financial fair play έχει στόχο να μειώσει τις πολύ μεγάλες ανισότητες. Και έτσι με το σύστημα αυτό, όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή, έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα σωστή κατεύθυνση. Τώρα, αυτό το οποίο αναφέραμε, δηλαδή η πτυχή της αλληλεγγύης ε, δεν ε, ισχύει στον ίδιο βαθμό. Και θέσατε το δάκλο επί των τύπων των ύλων και προτείνατε κάποιες λύσεις, ε, παραδείγματος χάρη το ερώτημα το εάν πρέπει να έχουμε άλλα μοντέλα αλληλεγγύης, τα τηλεοπτικά δικαιώματα, ένα ταμείο αλληλεγγύης, όλα αυτά είναι σωστά και χρήσιμα. Αλλά βεβαίως δεν νομίζω πως έχει φτάσει εκεί η συζήτηση και είναι λίγες οι δυνατότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γενικά ε, των ε, ευρωπαϊκών οργανισμών να δραστηριοποιηθούν. Δύο νούμερα τώρα. Το 2011 ε, στους συμμετέχοντες του Champions League 11-12 μοιράστηκαν 754 εκατομμύρια ευρώ και στο πλαίσιο της αλληλεγγύης 238 εκατομμύρια ευρώ. Βλέπετε το χάσμα. Οπότε πρέπει να πλησιάσουν αυτά τα δύο νούμερα μεταξύ τους. Ε, Βεβαίω ε, δεν σημαίνει πως θα χρηματοδοτηθούν έτσι όλες οι 600-700 επαγγελματικές ομάδες, αλλά ένα μεγαλύτερο ποσοστό. Τώρα, η UEFA συζητάει πολλές και διαφορετικές ε, προτάσεις, ακόμα και μια ε, συγχώνευση Europa League και Champions League. Εδώ πέρα θέλω να δώσω την εξή συμβουλή. Πρώτα απ' όλα πρέπει να συνεχίσουμε να παρατηρούμε με επικριτική διάθεση και κυρία Πακ, πρέπει να υπάρξει μια γενική και μόνιμη συζήτηση και ενασχόληση με το θέμα αυτό. Τώρα για τις ε, συστάσεις ε, υπάρχει κάτι το οποίο άμεσα μπορεί να γίνει περιορισμένο νομίζω. Με το άρθρο 165 της συνθήκης ε, η, συνθήκη, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να λάβει ρυθμιστικά μέτρα Οπότε, όπως ήδη υπόθηκε, πρέπει να προσφύγεται στην δημοσιότητα, αλλά βεβαίως και να συσσωρευτεί γνώση. Και νομίζω πως ε, και η Κομισιόν Συμβούλιο και η Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή ε, θα πρέπει να ασχοληθούν, να αποκτήσουν γνώση περί του θέματος, περί του ευρωπαϊκού αθλητισμού και ε, είτε μιλάμε για το οικονομικό πλαίσιο, το νομικό. Εδώ πέρα απαιτούνται περαιτέρω βήματα για να αποκτηθεί πρώτα απ' όλα μια βάση επί της οποίας μετά ίσως δραστηριοποιηθείτε. Δραστηριοποίηση τώρα. Τι σημαίνει αυτό. Κύριος μέσα δημοσιότητας, διάλογος, διάλογος με την ΟΕΦΑ και με τους άλλους οργανισμούς του αθλητισμού, αλλά επίσης κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία, να, υπόψη, ληφθούν υπόψη οι εθνικές ομοσπονδίες περισσότερο από ότι τώρα νομίζω ο διάλογος ε, με τα εθνικά κοινοβούλια έχει σημασία. Η ευρωπαϊκή πολιτική είναι νομίζω μια πολυεπίπεδη πολιτική και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τον αθλητισμό. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν ποιες δυνατότητες παρέμβασης υπάρχουν και στην Ευρώπη δεν έχουμε μόνο 27 κράτη-μέλη αλλά και 27 διαφορετικά αθλητικά συστήματα και το κάθε ένα προσπαθεί με το δικό του διαφορετικό τρόπο να προχωρήσει. Αλλά νομίζω πως τώρα πρέπει να ενισχυθεί ο διάλογος μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων και με τις Εθνικές Ομοσπονδίες για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επιτυχίες ειδικά ένα βασικό μεγάλο μέσο είναι οι κρατικές ενισχύσεις, ο ρόλος του κράτους φορολογικά μέτρα ή ελαφρύνσεις ε, για να υπάρξει βεβαίως και κάποια αλληλεγγύη αλλά βεβαίως και μια μείωση ίσως των μεγάλων δαπανών τώρα όσον αφορά τον βασικό ρόλο των διεθνών αθλητικών οργανισμών και έφτασα ίσως ε, στο θέματα των συναδέλφων. Εδώ πέρα θα μπορούσε το Κοινοβουλίο μαζί με Κομισιόν και Συμβουλίο ακριβώς επειδή έχει υπερεθνικό δίκαιο, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα σύστημα δικαίου, ε, ε, υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες στην Ευρώπη από ό,τι σε άλλες ε, υπήρους. Γιατί ακριβώς εδώ πέρα δραστηριοποιούνται πιο ελεύθερα οι διεθνείς αθλητικοί οργανισμοί και θα έπρεπε νομίζω να γίνει μια έκκληση για πιο δημοκρατική ε, λειτουργία. Και αυτό το οποίο είπε ο κ να δούμε και συγκεκριμένα άτομα, αλλά και διαρθρωτικά μέτρα. Το ερώτημα για ε, ελέγχους, δικλείδες ασφαλείας. Γιατί είναι τόσο αυστηρά η ιεραρχική η οργανισμοί του αθλητισμού. Πρέπει να υπάρχει και ένας μηχανισμός ελέγχου πέραν από αυτά τα οποία ε, είπαν οι συνάδελφοι. Εδώ πέρα νομίζω πως μπορεί να δραστηριοποιηθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε να κάνει τα παραπέρα βήματα και να μην ε, γίνει κάτι το στιγμιαίο, αλλά να υπάρξει μια διάρκεια. Σας ευχαριστώ κύριε Άντερσεν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους για τις πολύ ενδιαφέρουσες απαντήσεις που δώσατε σε πολύ δύσκολες ερωτήσεις που θα μπορούσαν να μας ε, ε, κρατήσουν όλη τη νύχτα εδώ για να συζητάμε και να απαντάμε σε αυτά τα θέματα. Επιτρέψτε μου να ε, προσεγγίσω ένα θέμα που δεν είναι στην ημερήσια διάταξη αλλά που το υπογράμμισαν πολλές ερωτήσεις. Τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη και τι μπορούν να κάνουν οι Ευρωπαίοι όταν έχουν ένα τεράστιο καθολικό φαινόμενο παγκοσμιοποιημένο για τον αθλητισμό ο οποίος εντάσσεται εκεί ε, έχει παγκοσμιοποιηθεί τρομακτικά τα τελευταία χρόνια. Οπότε οι συνάδελφοι στο Δανικό Ιστιντούτο Μελετών ε, υπέβαλαν μία παρουσίαση που έλεγε ότι υπάρχουν πολλά ε, προβλήματα, πολλές επιπτώσεις αρνητικές ότι αποχωρούν από την Ευρώπη, ότι πολλές αναδυόμενες οικονομίες και πολλές χώρες οι οποίες έχουν ε, τώρα μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση από ό,τι είχαν 150 χρόνια πριν θέλουν περισσότερη εξισορρόπηση στο θέμα του αθλητισμού, της ανανέωσης του αθλητισμού, των δικαιωμάτων των σχετικών και βλέπετε ότι η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική τώρα πια γιατί στα συνέδρια, στις ε, ε, διασκέψεις που γίνονται βλέπετε ότι οι πρόεδροι προέρχονται από μικρότερες χώρες, μικρότερες και βλέπετε ότι προέρχονται από μικρές ομάδες και έχουν ένα σύστημα ψηφοφορίας για ένα έθνος ενιαίο, κάτι το οποίο τους βοηθάει πάρα πολύ για να πετυχαίνουν τις πλειοψηφίες τις οποίες θέλουν, εκλέγουν προέδρους και αντιπροέδρους όπως το επιθυμούν, οι οποίοι είναι και πολύ ισχυροί. Ε, οι Ευρωπαίοι λοιπόν έχουν μια επιβραδυμένη θέση και επίσης είναι και ένα πρόβλημα με την ευρωπαϊκή αγορά. Υπάρχουν πάρα πολλά αθλήματα μέσα στην ευρωπαϊκή αγορά όπου κυριαρχούν ε, ορισμένα αθλήματα και υπάρχει ένα περιθώριο ελιγμού με ε, ελιγμού των πολιτικών οι οποίοι μπορούν να παρέμβουν ουσιαστικά. Ε, τι σημαίνει λοιπόν παγκοσμιοποίηση στην περίπτωσή μας. Η, ότι επίσης η μόρφωση και η επιμόρφωση είναι παγκοσμιοποιημένη. Ο καθένας θέλει να γίνει αρεστός. Ε, θέλει να γίνεται υποδεκτός με χαμόγελα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και όλοι αυτοί που ζουν μέσα σε έναν επαγγελματικό βίο πάρα πολύ καλά δομημένο ζητούν και απαιτούν το σεβασμό από τους συναδέλφους τους και αυτό έχει ένα ανθρώπινο στοιχείο, πολύ ανθρώπινο και ανακεφαλαιώνοντας θα ήθελα να πω ότι η φωνή της Ευρώπης είναι πολύ σημαντική. Μπορεί να υπάρχουν νομικά εμπόδια, αλλά είναι και πολιτικό αυτό το θέμα ταυτόχρονα και χαίρομαι που μπορώ να δηλώσω ότι ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρεί και εξελίσσεται προς τη σωστή κατεύθυνση. Και τώρα για να δούμε το σκέλος το αθλητικό πιο καλά, πιστεύω ότι πρέπει να πούμε ότι το στήσιμο των αγώνων και η διαφθορά μέσα στις ομοσπονδίες αλλά καθώς και το ντόπινγκ όλα αυτά είναι φαινόμενα τα οποία ε, είναι φαινόμενα παρέμβασης γιατί εμείς σεβόμαστε πάρα πολύ τους συνδέσμους. Για μας αντιπροσωπεύουν μια τεράστια αξία. Υπάρχει μια μεγάλη βιομηχανία η οποία παραμένει ανεξέλεγκτη. Έτσι παρουσιάζεται το θέμα σε εμά. Δεν υπάρχουν εξωτερικοί έλεγχοι επαρκής αλλά ούτε και εσωτερικοί έλεγχοι καθόλου. Και δεν γίνεται καμία μεταρρύθμιση, δεν έχει γίνει καμία μεταρρύθμιση ε, μετά από τόση πίεση για το, τους αρχηγούς, τους ηθήνοντες στο θέμα, των αγώνων είναι ένα θέμα γιατί ξαφνικά βρίσκονται με πάρα πολλά χρήματα στα χέρια τους και πρέπει να δράσουν και ε, όπως είπε ο Όσκαρ Γουάλντ, τα πάντα στα πάντα θα μπορούσα να αντισταθώ, στον πειρασμό όμως όχι. Ε, Βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση λοιπόν και υπάρχουν τα δίκτυα. Τα δίκτυα μπορούν να παράγουν έλεγχο εξωτερικό που να είναι επαρκής αν ακούσετε τη σημαντική συζήτηση που είχαμε σήμερα, το στοιχείο αυτό είναι πραγματικά ενθαρρυντικό. Το 2006 θυμηθείτε ότι είχε υπάρξει μια καθολική συστηματοποίηση σε διεθνές επίπεδο, πολύ περισσότερο διεθνές, και είχαμε προτείνει ένα θεσμό που θα αντιστοιχούσε με την εταιρεία anti-doping, η οποία θα ήταν μια εταιρεία κατά της διαφθοράς και του στισίματος των αγώνων, όπως υπάρχει εταιρεία αντιντόπινγκ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τεράστια επιθυμία δαπάνησης χρημάτων για την ώρα και γι' αυτό νομίζω ότι υπάρχει δισταγμός και γενικευμένος δισταγμός. Άλλαξα λοιπόν την πρόταση υπό το φως των όσων λέμε είπα ότι πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε με σαφήνεια ανταλλαγή πληροφόρησης και οι υπηρεσίες των αγώνων και του αθλητισμού θα πρέπει να έχουν μία σφραγίδα ποιότητας την οποία να την ε, χρησιμοποιούν μετά από έλεγχο των κυβερνήσεων, μετά από έλεγχο των πάντων. Βέβαια, ο καλύτερος τρόπος πιστεύω να έχει κανείς ε, αξιοπιστία ε, είναι να την βρίσκει από αλλού την αξιοπιστία, δηλαδή να μην την ζητάει από τον εαυτό του, να είναι εξωτερική η αναγνώριση. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα διεθνές όργανο με ελεγκτές ε, διεθνούς χαρακτήρα που θα μπορεί να εγγυάται τον την εντιμότητα ενός αγώνα και να βάζει τη σφραγίδα του. Και νομίζω ότι αν κοιτάξουμε προς αυτή την κατεύθυνση, πραγματικά όλα αυτά μπορούν να γίνουν σε θελούσια βάση. Και ας προσθέσω και το εξή. Για τον νόμο δεν είμαι νομικός, αλλά πρέπει να πω ότι σε ό,τι αφορά τον νόμο, ε, οι περισσότερες αθλητικές οργανώσεις βρίσκονται στην Ελβετία. Η Ελβετία έχει ε, πληγεί και επηρεαστεί πάρα πολύ από το πρόσφατο τη σκάνδαλο της FIFA και την απασχολεί το θέμα των διεθνών οργανώσεων αθλητισμού. Είναι και ένα πολιτικό θέμα. Έτσι βλέπει κανείς ε, πώς μπορεί να αντιμετωπίσει τα διεθνή θέματα που είναι, χαρακτηρίζονται από μεγάλη ασάφεια και ε, πώς μπορεί να αλλάξει νομοθεσία. Ε, εγώ μιλούσα για αυτά τα προβλήματα και πιστεύω ότι, από το δύο, ότι μπορεί κάτι να αλλάξει μέσω της Ελβετίας. Ότι ήδη από το 2006 που είχαμε μια συζήτηση η επιθυμία αλλαγή στην Ελβετία υπάρχει. Η Ελβετία αναγνωρίζει ότι ακριβώς επειδή υπάρχει πολιτική πίεση και πίεση από τα μίντια και από την κοινή γνώμη αποφάσισε όχι, η Ελβετία ε, ότι δεν θα δώσει πλήρη ελευθερία στους συνδέσμους ε, για να χρησιμοποιούν και να καταχρώνται των προνομίων τους. Ε, βεβαίως δεν άλλαξε τίποτα στην ελβετική νομοθεσία για την ώρα, αλλά υπάρχει πιθανότητα να γίνει αλλαγή στο μέλλον και ε, σύντομα μπορώ να πω ότι ο συντονισμός σε διεθνές επίπεδο είναι απόλυτα αναγκαίος και πάρα πολλές διεθνείς ομάδες ε, δείχνουν σκεπτικισμό όταν ε, ακούν ε, κάτι τέτοιο. Ωστόσο άλλες είναι θετικές και θέλουν να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών, χρειάζονται πόροι για να υπάρχει παροχή υπηρεσιών και να υπάρχει βοήθεια και στήριξη στις διεθνείς ομοσπονδίες. Ευχαριστώ. Να προσθέσω σε αυτό το οποίο είπε ο από την Europol πως ε, καλά σας είχα καταλάβει. Δεν νομίζω πως κάποιος από μας ε, θα έλεγε σε κάποιον νέο πως ε, που μπλέξει κάτι τέτοιο πως θα τον επιβαρύνει σε ολόκληρη τη ζωή του. Αλλά όταν λέμε μηδενική ανοχή, ε, μιλάμε για επαγγελματισμό. Αυτό εννοούμε, όχι ε, όταν κάποιο ε, κάποιος νέος αθλητής μπλέξει σε μια τέτοια υπόθεση. Ε, ε, εκεί πέρα εντάξει υπάρχει και επίκαια. Έτσι, για, να συνεννοούμαστε. Αυτό, και αυτό με τη σφραγίδα που είπατε, καλή είναι, ίσως θα πρέπει να το σκεφτούμε. Δυστυχώ είχες δίκιο, Σαντιάγκο. Το μιλάμε για ελβετικό δίκαιο, το οποίο αμφισβητείται και στην Ελβετία, έχεις δίκαιο τις νέες δυνατότητες εφευρημάτων, όπως είπες. Και μετά λένε ότι τους ανάγκασαν να το αποσύρουν. γιατί, ποιος τους ανάγκασε. Ποιος μας ανάγκασε να μην, να μην το δεχτούμε αυτό. Θα το δούμε. Λοιπόν, στον αθλητισμό που φαίνεται πως ε, η παγκοσμιοποίηση φέρνει μεγάλους, έχει μεγάλους πειρασμούς και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τις περιορισμένες δυνατότητες μας. Λοιπόν, έχουμε κάποιον από την Κομισιόν εδώ πέρα. Ο Τζεν Λούκα Μέντε. Έχετε το λόγο. Θέλεις, θέλεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε. Πολλά θέματα εθίγησαν σε ό,τι αφορά το ζήτημα του οικονομικού αγωνίζεστε είναι κάτι το οποίο ε, μας μίλησε ο ε, προσκεκλημένος μας ακούσαμε ενδιαφέροντα πράγματα υπάρχουν κάποια σχέδια αναφορικά με προπαρασκευαστικές δράσεις ε, για τον αθλητισμό ε, θα μπορούσα να σας ε, παρέσχω μια σχετική ενημέρωση. Στις αρχές του 2013 θα έχουμε μια παρουσίαση που θα γίνει για το ζήτημα αυτό. Και τώρα θα ήθελα να επικεντρώσω την παρέμβασή μου το ζήτημα του match fixing, δηλαδή της, ε, των στημένων αγώνων. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η νομοθεσία δυστυχώς ε, ε, Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, αλλά υπάρχουν ορισμένα θέματα που μπορούν να βελτιωθούν σε κάποιου τομεί και να μιλήσω για το, ένα ζήτημα το οποίο δεν εθίγει, δηλαδή το θέμα της πρόληψης. Όλοι οι εμπλεκόμενοι συμφωνούν ότι η πρόληψη είναι σημαντική για την, το ε, θέμα της ε, στο θέμα μάλλον των στοιχημάτων των αγώνων. Και εδώ ξέρουμε ότι εμπλέκονται οι προπονητές, ε, παίκτες ε, και ούτω καθεξής και εμείς επιλέξαμε 7 προγράμματα στο πλαίσιο της προπαρασκευαστικής δράσης. Θα ξεκινήσουμε την επόμενη χρονιά να τις εφαρμόζουμε και να προωθήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές. Ορισμένα πράγματα έχουν γίνει σε εθνικό επίπεδο, σε ορισμένα αθλήματα, όχι σε όλα. Θέλουμε λοιπόν να συνδυάσουμε όλες αυτές τις προσπάθειες που έχουμε στην διάθεσή μας και συζητήσαμε το πρόβλημα στο ζήτημα της ε, εκπαίδευσης, ε, κατάρτισης, ε, κάτι το οποίο θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση με τα μέσα που έχει και να προωθήσει τις, τις προσπάθειές μας που έχουμε ξεκινήσει να εφαρμόζουμε τώρα ό,τι αφορά το άρθρο 165 της συνθήκης δεν μπορούμε να, να το χρησιμοποιήσουμε και να μας βοηθήσει στις προσπάθειές μας. Ο κύριος Φίσας, ε, Φίζας ε, ε, ε, συνέταξε μία έκθεση και η μελέτη έχει δημοσιευτεί και αφορά στο ότι κάποια κράτη-μέλη έχουν ε, την ε, νομοθεσία την οποία και εφαρμόζουν. Ορισμένα όμως κράτη δεν έχουν το απαραίτητα ε, νομοθεσία για την καταπολέμηση της διαφθοράς έχουν αναλυφθεί κάποιες δραστηριότητες Κάποια κράτη έχουν αναλάβει την ε, δικαστική δίεξη και ίσως ε, μορισμένη νομοθεσία που φυσικά χρειάζεται μια διαδικασία μακροχρόνια μπορεί να βοηθήσει μεν, αλλά αυτό που απαιτείται είναι η συνεργασία και πάντα σε σχέση με την νομοθεσία όλοι γνωρίζουμε ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης ε, διαπραγματεύεται μελλοντική σύμβαση για το θέμα των, ε, των στημένων παιχνιδιών. Το τρίτο σημείο είναι η συνεργασία. Αυτό υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη και περισσότερη συνεργασία όλων των ε, εμπλεκομένων, καταπολέμηση του στισίματος των αγώνων. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι παίζουν έχουν ο καθένα σημαντικό να διαματήσουν όπως η επιβολή της ε, νομοθεσίας, συνεργασία με την Eurojust ε, την... Ε, και άλλου οργανισμού. Επίσης να αναφέρω ότι η Κομισιόν στις 23 Οκτωβρίου έκανε ένα πρόγραμμα δράσης για τα στοιχήματα τι μπορούμε να κάνουμε για περαιτέρω συνεργασία. Υπάρχει μια, εμπειρογνω... μια ομάδα εμπειρογνωμόνων ε, που ανταλλάσσουν προφορίες ε, σε διάφορα ζητήματα και ένα από αυτά τα ζητήματα είναι η προστασία της ακεραιότητας ε, των αθλημάτων και ένα άλλο σημείο του πρόγραμματος δράσης είναι οι συστάσεις Κομισιόν το 2014 θα εγκρίνει τις βέλτιστες πρακτικές και στο τι μπορούμε να κάνουμε για την ε, καλύτερη συνεργασία της πρόληψης και της καταπολέμησης ε, του στισίματος των παιχνιδιών και κάποια παραδείγματα που θα θέλαμε να εφαρμοστούν στον τομέα της απαγόρευσης στοιχημάτων ε, που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο, σε κάποιες αθλητικές ενώσεις, πώς επιβάλλονται, ιδιαίτερα σε διασυνοριακό επίπεδο και επίσης πώς μπορούμε να ανταλλάσσουμε προφορίες ε, αναφορικά με υποπτά στοιχήματα. Όταν υπάρχουν λοιπόν υποψίες ε, τότε θα πρέπει να ανταλλάσσονται οι πληροφορίες. Ε, θέλουμε να εξετάσουμε περαιτέρω το θέμα σε εθνικό επίπεδο και σε διασυνοριακό επίπεδο για να παρέχουμε βοήθεια και αρρωγή σε αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Βλέπουμε πως η Κομισιόν παρά το ότι ε, προσφάτως αποκτήσαμε κάτι αρμοδιότητε σε αυτό το τομέα έχει ήδη κινητοποιηθεί. Χαιρόμαστε γι' αυτό, το είχαμε ζητήσει και θεωρώ πως είναι στο σωστό δρόμο και θεωρώ πως πρέπει στον ε, τομέα αυτόν και σε άλλους τομέες όπου έχουμε μόνο επικουρικές αρμοδιότητες να προσπαθήσουμε να μάθουμε ένας από τον άλλον. έτσι ώστε να υπάρξει κάποια εναρμόνιση. Για ζητήματα, όπως είπα, στα οποία έχουμε κάποιες επικουρικές αρμοδιότητες. Αναφερθήκατε σε κάποια οργανωμένη σιωπή, η οποία σπάει, άρα πρέπει να μιλήσουμε δυνατότερα και όχι μόνο μία φορά, αλλά σε τακτά χρονικά διαστήματα να επαναφέρουμε το θέμα. Γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς, ποιος θα το κάνει. Έχουμε κάποιες αρμοδιότητες. Ξέρουμε πως ε, πρέπει να διατηρούμε το θόρυβο γύρω από αυτό το θέμα και τις ε, ηθικές επιφυλάξεις που υπάρχουν. Ευχαριστώ λοιπόν ιδιαίτερα τους τρεις ειδικού μας. Ο τρίτος έλειπε. Αλλά εντάξει δεν θα τον καθίσουμε σκαμνή. Και χάρηκα για το ότι συμφωνούμε σε πολλά πράγματα και μάθαμε από εσά που ε, είναι οι δυνατότητες δράσης. Θα αναζητήσουμε διάλογο με την ΟΕΦΑ Ευχαριστώ και επίσης και την Κομισιόν, διαφωτιστικά αυτά τα οποία μας είπατε. Και στο πλαίσιο αυτό να ευχαριστήσω την βιβλιοθήκη μας που έκανε εξαιρετική έρευνα. Αν δεν το έχετε, να το πάρετε γιατί είναι πραγματικά... Ε, δεν είναι πολλά, αλλά είναι διαφωτιστικά. Μας δίνει δυνατότητες για την καθημερινή μας εργασία. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που ήρθαν. Ευχαριστώ και τους εμπειρογνώμονες. Ολοκληρώθηκε ε, η συνάντηση. Παρακαλώ να υιοθετήσετε τις συστάσεις των συντονιστών. Ωραία, σημείο 12, διάφορα, υποθέτω πως δεν έχετε να πείτε τίποτα άλλο. Επόμενη συνεδρίαση 23-24 Ιανουαρίου, σκεφτείτε επίση την προθεσμία των τροπολογιών ε, για την έκθεση του Μπόρις είναι Τετάρτη του Στρασβούργου. Πέμπτη, πέμπτη, 17. Μάλιστα, μην το ξεχάσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους παρόντες, ευχαριστώ τους διερμηνείς. Καλά Χριστούγεννα και σε αυτούς και οπωσδήποτε ευτυχές το νέο έτος. Δύσκολα πράγματα και το επόμενο έτος πολλά λεφτά και πολλά προγράμματα πρέπει να δώσουμε. Λοιπόν, ας ε, κάνουμε και λίγο έτσι Χριστούγεννα με την ησυχία μας. Ευχαριστώ και γεια σας.